Um, Ας ξεκινήσουμε φίλοι μας. Κάπου χάθηκε η πρόεδρος. Δεν ξέρω πού είναι ο πρόεδρος. Uh, και δεν είμαστε και πολλοί εδώ. Θα καταφθάσουν όμως αργότερα και οι υπόλοιποι. Δεν είμαστε πολλοί, οπότε τα σχόλιά μου θα είναι και σύντομα. Χαίρομαι που διεξάγεται αυτή η πρώτη μήνυ ακρόαση στα πλαίσια της, νομοθ... της έκθεσης πρωτοβουλίας Επιτροπής ε, Βολτικών Ελευθεριών, ιδίας πρωτοβουλίας για την εποπτεία και την επιβολή του κράτους δικαίου και των θεμελιών δικαιωμάτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. που θεωρώ το σύμφωνο δημοκρατικής διακυβέρνησης ότι αυτός ο τίτλος ταιριάζει καλύτερα, είναι πιο συμπαγής. Ε, είναι η πρώτη ακρόαση που ελπίζω που θα, τελικά θα καταλήξει να είναι μια μήνυ σειρά ακροάσεων. Θα έχουν περισσότερες τον επόμενο χρόνο. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε σε κάποια τα ψηφίσματα ότι θα ετοιμάσει μια πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου ζητώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποβάλει προτάσεις για ένα σχετικό μηχανισμό διότι όλοι βλέπουν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλλειψη μέσων ούτω ώστε να μπορεί πραγματικά να επιβάλλει την δημοκρατική διακυβέρνηση, θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Έχουμε κάποια νομοθετικά μέσα τα οποία είναι περιορισμένα και πολύ συγκεκριμένα και απ' την άλλη έχουν την, το πυρηνικό όπλο, το άρθρο 7. Α, καλημέρα. Νόμιζα ότι θα έρθεις τρέχοντας. Θα είμαι πολύ σύντομη λοιπόν. Χρειαζόμαστε κάτι για να καλύψουμε το κενό διότι έχουμε δύσκολες συζητήσεις τώρα για συγκεκριμένες χώρες ή υποβάλλουμε κοινοβουλευτικά ερωτήματα και δεν οδηγούν αυτά σε κάποια δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλη λέει, κοιτάξτε δεν έχουμε τα μέσα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Οπότε με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Ήδη έγιναν κάποιες αρχικές συνεδριάσεις των σκιωδών και αποφασίσαμε να τεμαχίσουμε σε τμήματα την έκθεση και κάθε σκιώδης εισηγητής θα είναι υπεύθυνο για την σύνταξη ενός τμήματος ούτως ώστε θα έχουμε ένα κοινό εγχειρήμα, κοινή προσπάθεια και είναι κάτι που θα λάβει μορφή τους επόμενους μήνες. Δεν είναι όπως όταν έχουμε ένα θέμα, ετοιμάζει ο εισηγητής ένα σχέδιο κειμένο και μετά ψηφίζουμε και μετά έχουμε 50% των ψήφων συνένα, όχι. Εδώ θα το οικοδομήσουμε αυτό μαζί και στη συζήτηση θα διαμορφωθούν διάφορες ιδέες σχετικά με την πορεία μας. Ο μηχανισμός που θα αναπτύξουμε θα ισχύει όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμπεριλαμβάνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ιδίας, ε, διότι αν πούμε ότι περιμένουμε τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε κάποια πρότυπα και εμείς σαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο, αυτό είναι σίγουρο. Σήμερα λοιπόν θα εστιάσουμε τη συζήτηση επί του θέματος των μεθόδων και των δικτών. Διότι όταν μιλάμε για δημοκρατία κάτω δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα, χρειαζόμαστε δείκτες για να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δείκτες στα κάτι μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα που να συζητήσουμε, διότι η αρχική αντίδραση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Επιτρόπου Τίμερμαν ήταν η εξή. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοια μέσα, διότι δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε, να ποσοτικοποιήσουμε τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Συνεπώ, αυτό το εργαλείο δεν θα λειτουργήσει. Νομίζω ότι είναι αυτή η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να αποδείξουμε ότι κάνει λάθο και να επεξεργαστούμε την κατάρτιση αυτή των δικτών. Αυτά θα ήθελα να πω εν είδη εισαγωγής. Και τώρα δίνω τη σκητάλη στον Πρόεδρο που θα κάνει την πραγματική έναρξη της ε, συνεδρίας σας. Συγγνώμη, Σοφή, που ζητώ συγγνώμη. Ασυνήθιστη καθυστέρησή μου. Έπρεπε να πάω σε τρεις διαφορετικούς ορόφους να βρω την κάρτα ψηφοφορίας και πάντα αυτό σας λέω να κάνετε εσείς. Και όπως ξέρετε έχω και πρόβλημα με τον αστράγαλό μου και δεν περπατούσα γρήγορα. Αυτή είναι η περίπλοκη δικαιολογία μου, ζητώ συγγνώμη. Αυτά. Ξανά συγγνώμη. Ευχαριστώ Σοφή που ξεκίνησες τη συνεδρίαση. Περιτός εγώ πιστεύω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Με την κυρία Μίσιο. Μίχου. Μίχου. Λοιπόν, ξεκινήστε και είστε ευπρόσδεκτοι. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα και πάντα χαίρομαι και απολαμβάνω να βρίσκομαι ε, υπό την προηγούμενη θέση μου ως ε, ανακριτής διευθυντρία της ε, Γενικής Διεύθυνσης και χαίρομαι γιατί έχω λίγο πολύ τις ίδιες ε, ευθύνες και αρμοδιότητες στη Γενική Διεύθυνση. Κάποιες από αυτές έχουν να κάνουν με θέματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων και στην παρούσα φάση λοιπόν ασχολούμαι με όλα αυτά τα μέτρα μετανάσταση, ασφάλειας, κράτος δικαίου και γι' αυτό λοιπόν έχω έρθει εδώ. Σοφή, δεν ε, φαντάζομαι να περιμένεις να αντιταχθώ στον αντιπρόεδρο, στον πρώτο αντιπρόεδρο, αλλά να διαβεβαιώσω όλους τους βουλευτές mm. ότι εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ενδεχομένω να μην έχουμε προτείνει νέους μηχανισμούς, νέους δείκτες, όχι κάτι παραπάνω από αυτά που είχαμε ως τώρα τουλάχιστον, αλλά νομίζω ότι βάσει των όσων έχουμε στα χέρια μας καταφέραμε να πετύχουμε πολλά. Και θεωρούμε Ακούσατε άλλωστε και τον πρώτο αντιπρόεδρο αλλά και την επιτρεπό Γιούρεβα τι είπαν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας αρκούν για να επιτελέσουμε το έργο μας. Επίσης, εκτιμούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να μας χορηγήσετε κάποια στοιχεία. Η Επιτροπή δεν θα είναι αυτή που θα αποδράσει από το να συμμετάσχει, αν θέλετε, στο εγχείρημα αυτό, στην ε, άσκηση αυτή. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θεμελιώδη δικαιώματα και στο κρατός δικαίου. Και γι' αυτό λοιπόν έχει θέσει τον πρώτο Πρόεδρο αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα, στα χρόνια, με, με την παράδοση του χρόνου, έχει εργαστεί σκληρά για να καταρτήσει ένα πρόγραμμα. Και ήρθα λοιπόν για να σας μιλήσω για το scoreboard, για το πώς χρησιμοποιούμε την ε, εξουσία δράσης επί όταν βλέπουμε ε, ότι τα κράτη-μέλη προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας και εξέτασης και επίσης, όπως είπε ο κύριος Τίμερμανς, γνωρίζουμε ότι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί μια καθημερινή εργασία και θα πρέπει να διατρέχει αυτό όλες τις πολιτικές από τη φάση της, ε, του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της κατάρτισης μέχρι και την φάση της υλοποίησης. Τι κάνουμε λοιπόν, προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνεται επί τόπου, προκειμένου να ξέρουμε και να μπορούμε να δράσουμε αναλόγως. Και θα ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για μεθοδούς ε, αξιολόγησης ε, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου στα κρατη και ιδιαίτερα για τις εμπειρίες που έχουμε εμείς στον τομέα αυτό. Θα επικεντρωθώ λοιπόν τώρα συνοπτικά, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε και πολλές ερωτήσεις, θα επικεντρωθώ λοιπόν σε τρία βασικά εργαλεία. Το Ευρωπαϊκό Σκορμπορ για την Δικαιοσύνη, ο Μηχανισμός για το Κράτος Δικαίου και ο, η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της χάρτας. Έχουμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ασφαλώς. Έχουμε και το μηχανισμό επιβεβαίωση συνεργασίας, ο οποίο είχε συμφωνηθεί στη φάση των προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Και εκ έχουμε βέβαια, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση εμ, διαφθοράς του 2014 και επίσης έχουμε και τις στοχευμένες δράσεις τις οποίες προσπαθούμε να, με τις οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους εθνικούς ε, θεσμούς για το κράτος δικαίου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση του δικαστικού, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την μεταρρύθμιση της ε, δημόσιας διοίκησης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση και το έχουμε κάνει σε διάφορες περιστάσεις όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η σχετική υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων θα γίνει και μια παρουσίαση πιο μετά. Παρέχει αρρωγή και εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα. Συλλέγουν λοιπόν και μας παρέχουν ε, αντικειμενικές ε, πληροφορίες και τα αποτελέσματα της εποπτείας και αυτά όλα χρησιμοποιούνται στην ε, εργασία και των θεσμικών οργάνων και της Ένωσης και των κρατών μελών. Τέλος. Να μην ξεχνάμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες που κατοχυρώνονται στη συνθήκη στο scoreboard. Ξέρετε ότι έχω έρθει να σας παρουσιάσω τα σχετικά αποτελέσματα για την δικαιοσύνη για φέτος. Έχουμε έναν ε, καλό μηχανισμό που σχετίζεται και με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και Οικονομικής Προσαρμογής. Τρία έτη μόνο χρησιμοποιείται αυτός ο μηχανισμός, είναι σχετικά καινούριο. Και μέσα από τον πίνακα αυτό, το scoreboard αυτό, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε στενά τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα το δικαστικό στα κράτη-μέλη. Κάθε χρόνο δε, το Συμβούλιο εγκρίνει βάση του πίνακα αυτού τις συγκεκριμένες συστάσεις βάση και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. υποστηρίζει την διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμένου Και είναι πραγματικά απαραίτητος μηχανισμός, και αυτό το βλέπουμε κάθε έτος, προκειμένου να γίνεται μια συγκριτική ανάλυση, μια επισκόπηση για το πώς ε, λειτουργούν οι μεταρρυθμίσεις του αστικού, εμπορικού και δικαστικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Γίνεται και μια πολύ προσεκτική ε, ενδελεχής ανάλυση και αυτό πρέπει να γίνεται από όλους και εμείς ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Scoreboard για τη δικαιοσύνη συμπληρώνουμε τα στοιχεία αυτά με μια πιο ενδελεχή ανάλυση. Φέτος δε θα είναι λεπτομερέστερη η ανάλυση σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του συστήματος. Άρα κάθε χρόνο προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε τον πίνακα αυτό και με νέα στοιχεία. Θα ήθελα όμως να τονίσω και ιδιαίτερα τη διάσταση της συγκρισιμότητας των στοιχείων. Κάθε χρόνο αυτό αποτελεί πολύ καλή πηγή ανάλυσης. Προσπαθούμε επίσης να τα επαληθεύουμε τα στοιχεία αυτά. Όταν μιλάμε για δικαστικά συστήματα, ασφαλώς θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε για τα δεδομένα που έχουμε, τόσο πιο σίγουροι είμαστε για τα αποδεκτικά στοιχεία όταν χρειαστεί να αναλάβουμε δράση. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το δικαστικό. Με τη με τη Eurostat ε, και με πολλές άλλες ε, αρχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Να σας μιλήσω λοιπόν ότι ο μηχανισμός ε, για το κράτος δικαίου δεν είναι μηχανισμός παρακολούθησης για μας, αλλά ένας μηχανισμός για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιπτώσεις που θεωρείται ενδεχομένως ότι θα αποτελούσαν κίνδυνο για το κράτος δικαίου. Η Επίτροπος Γιούροβα και ο πρώτος αντιπρόεδρος ασφαλώς εξήγησαν και μάλιστα η Επίτροπος Γιούρεβα το έκανε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί όπου υπάρχει σαφής ένδειξη συστηματικής απειλής του κράτους δικαίου σε ένα κράτος. Ιδιαίτερα μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με διαδικασία επιπαραβάση και επί... όταν οι εθνικοί μηχανισμοί δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Το πλαίσιο λοιπόν ζητά μια αντικειμενική και λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης και αυτό συνδέεται με αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως. Χρειάζεται να έχουμε γνώση και επίγνωση συγκεκριμένων καταστάσεων για το κράτος δικαίου σε κάθε κράτος μέλος και αναζητούμε ε, την εμπειρογνωμοσύνη και εξωτερικών ε, σωμάτων, όπως η Υπηρεσία τα Δικαιώματα, η Επιτροπή της Νίκαιας, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ανάλυση της ε, προκειμένης κατάστασης κάθε φορά. Και πιστεύουμε ότι το κράτος δικαίου σε κάθε κράτος μέλος δεν μπορεί να ποσοτικοποιείται μηχανικά με δείκτες. Χρειάζεται μία ποιοτική εξέταση πάντα της κατάστασης και αξιολόγηση. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ετήσια έκθεση. Από το 2000 από ό,τι είδατε. Παρουσιάζει λοιπόν τις αξίες μιας ελεύθερης και περιεκτικής ε, ανοιχτής κοινωνίας και νομίζω ότι όλοι έχουμε ευθύνη να προωθούμε τις αρχές αυτές καθημερινά, στις καθημερινές μας δράσεις και ενέργειες. Η αιτήσια, λοιπόν έκθεση καταγράφει το πώς εφαρμόζονται οι χάρτες αυτές, αυτοί, από τα θεσμικά όργανα, από τα κράτη-μέλη, αποτελώντας τη βάση εφαρμογής των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη χάρτα και φέτος για πρώτη φορά υπάρχει και ένα νέο τμήμα για ένα θέμα το οποίο ανακύπτει όλο και πιο έντονα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την εμπειρία που είχαμε λοιπόν από όλα αυτά τα μέσα, από, όλα αυτές, από όλες αυτές τις εκθέσεις τα τελευταία χρόνια, είναι απόλυτα πεπισμένη πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της δημοκρατίας των θεμελιωτών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου είναι συχνά πολύ σύνθετα και πάντα, πάντα όπως είπα και προηγουμένως, προαπαιτούν μια ποιοτική σε βάθος ανάλυση για τους υφιστάμενους ε, κανόνες και τις υφιστάμενες πρακτικές στα άλλα κράτη-μέλη το επίπεδο των της των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου δεν μπορούν να μετρηθούν με τη μεζούρα. Δεν μπορεί να υπάρξει μηχανική ποσοτικοποίηση με άκαμπτους ε, Και δεν θα ήθελα να σας παρουσιάσω απαραίτητα τον μηχανισμό επαλήθευσης της συνεργασίας για να μην μακρηγορήσω, να απαντήσω καλύτερα στις ερωτήσεις σας. Αλλά να ξέρετε ότι παρακολουθούμε στενά την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Διοργανώνουμε και αποστολές στα κρατη αυτά και δημοσιεύουμε εκθέσει κάθε χρόνο. Αυτό το κάνουμε με πολλά αντικειμενικά στοιχεία με δείκτες που υποδεικνύουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στο οποίο δίνει στοιχεία ο πίνακας επιδόσεων αυτό το Ευρωπαϊκό Scoreboard για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου, τον οποίο παρακολουθούμε στενά, οι διαδικασίες επί παραβάση, βάσει των συνθήκων και όλες οι άλλες εκθέσεις, όλα αυτά θεωρούμε ότι μας δίνουν ένα πλωστάσιο με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει στο παρελθόν. Να κλείσω λέγοντας ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που καταβάλει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας για να υποστηρίξει τις θεμελιώδεις αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα επί των οποίων βασίζεται η Ένωση. Θα, παρακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη δουλειά σας και την ε, πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ να απαντήσω σε όποια ερώτηση έχετε. Ευχαριστώ κυρία Μίχου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο ε, Γκάμπριελ ε, Τόγενμπουργκ, που είναι από τον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων ε, νομικός σύμβουλος. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά ερχόμαστε εδώ, αλλά μπορεί να φαίνεται αυτό αντιφατικό. Αν χρειάζεται μηχανισμός για την προστασία του άρθρου 2. Είναι πολιτικής φύσεως αυτή η απόφαση Uh, ε, και είναι κάτι που αφορά ένα εξωτερικό εμπειρογνώμονα, οπότε αναρωτιέται κανείς τι δουλειά έχει ο οργανισμός της Βιέννης να έρχεται στις Βρυξέλλες να το συζητάει. Η απάντηση θα έρθει στο έγγραφο πολιτικής ε, και των τριών θεσμικών οργάνων που συμφωνούν επί δύο αρχών. Η πρώτη λέγει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση και το δεύτερο είναι ότι είπαν όλα τα θεσμικά όργανα ότι θα πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι και στοιχεία. Σήμερα τι θέλω να κάνω μαζί σας, να μοιραστώ ε, δύο εμπειρίες του οργανισμού μας και να κάνω και μία πρόταση. Ποιες είναι οι δύο εμπειρίες που είχαμε. Για τους δείκτες, αφορά η πρώτη και η δεύτερη αφορά πώς αντιλαμβανόμαστε την ε, Ένωση ως πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Για τους δείκτες λοιπόν χρησιμοποιούμε το SPO ε, που είναι μια έννοια του ΟΗΕ. Δηλαδή όχι μόνο να δούμε τι νομοθεσία υπάρχει, αυτή είναι η δομημένη, η διαρθρωμένη προσέγγιση, αλλά να δούμε και τι συγκεκριμένες πολιτικές προσπάθειες καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Στη διαδικασία της εκπόνησης, δηλαδή της εκτέλεσης και επίσης είμαστε φιλόδοξοι θέλουμε να καταλάβουμε κατά πόσο αυτές οι πολιτικές προσπάθειες πιάνουν τόπο και επιφέρουν καμιά αλλαγή στον πραγματικό κόσμο και στους πραγματικούς ανθρώπους, στις ζωές τους. Αυτό λοιπόν θέλουμε, να έχουμε αυτούς τους ε, δείκτες του ΟΗΕ ε, που ε, εξετάζει τις δομές, τις διαδικασίες και το αποτέλεσμα στα δικαιώματα των παιδιών, ε, στα ε, δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα τομέα που είναι η ένταξη των Ρωμά. Γιατί στην περίπτωση αυτή ήδη υπάρχει ένα σύστημα αναφοράς Ξέρετε ότι υπάρχει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταθέτουν στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά και στη συνέχεια το 2013 ε, υπήρξε κατάλογος ε, εκτενής και λεπτομερής ε, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό που έλειπε όμως ήταν κάποιες επιδόσεις μετρήσιμες ή που να έχουν μετρηθεί. Και εδώ μπαίνει ο δικός μας οργανισμός θεμελιωδών ελευθεριών, έκανε μια ομάδα εργασίας με 18 κράτη-μέλη και πρόσφατα καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί των δικτών με τα κράτη-μέλη. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία, διότι βεβαίως είναι δύσκολη η υπόθεση και θέλει να ε, κάνουν μια προσπάθεια και τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τα πρόκειται για ε, μη νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά το λεγόμενο soft law, εθελοντικής εφαρμογής. Όταν έχουν δείκτες, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται και δεν μπορούν να υπεκφεύγουν με διάφορες δηλώσεις ότι έλαβα το τάδε μέτρο και το δίνα μέτρο. Όχι, είναι ένας κορσές και πρέπει να ε, δεσμεύεσαι να υλοποιείς κάποιους στόχους, να συμπληρώνεις κάποια ε, ερωτηματολόγια, κάποιους πίνακες, templates κτλ. Είναι δύσκολο λοιπόν να συμφωνήσει κανείς σε δεσμευτικούς δείκτες που στη συνέχεια θα το κάνουν να λογοδοτεί επί συγκεκριμένων δράσεων, αλλά όχι αδύνατο. 18 ε, κράτη-μέλη συμφώνησαν λοιπόν και τώρα ε, αυτός ο πίνακας είναι το εργαλείο με το οποίο κάνουν τις αναφορές τους όλα τα κράτη-μέλη. Και υπήρχε αυτή η ανάγκη ε, δικτών, αλλιώς δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Είναι εύκολο να λέμε να έχουν πρόσβαση τα παιδιά των Ρωμά στη μόρφωση και στο σχολείο. Ωραία. Από εκεί και πέρα αυτό μου τι σημαίνει. Να έχουν εγγραφεί στο σχολείο. Να πηγαίνουν στο μάθημα. Ε, να μην έχουν απουσίες σημαίνει να πάρουν και ενδεικτικό ή απολυτήριο ε, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Τι σημαίνει πρόσβαση στη παιδεία γενικά και αόριστα όχι. Με δείκτες και με μετρήσιμα στοιχεία. Για να κλείσω λίγο αυτό το θέμα των δικτών θα ήθελα να πω το εξής για τις νομικές ε, ρυθμίσεις αυτό είναι εύκολο. Αυτό που ε, ε, είναι δύσκολο είναι να συμφωνήσουν για τις διαδικασίες για να ανταποκριθούν σε αυτό το νόμο. Έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα με τρεις χώρες, Ολλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία και ο στόχος ήταν. Ωραία, συμφωνήσαμε για τους δείκτες. Μπορούμε να βάλουμε στοιχεία που έχουμε ήδη από τους ελέγχους. Γιατί αυτή είναι η κλασική αντίρρηση, ότι δεν χρειαζόμαστε νέα εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης, έχουμε στοιχεία. Ωραία, τα στοιχεία που έχουμε μπορούμε να τα παντρέψουμε, να τα συνδυάσουμε με ε, αυτούς τους δείκτες του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ κτλ. Καταλήξαμε λοιπόν ε, στα εγκλήματα μίσου, στη ε, πρόσβαση ε, στη δικαιοσύνη και τις διακρίσεις και την ανεξαρτησία των, δικαστικών, των δικαστικών σωμάτων. Σε αυτά τα τρία θέματα είναι εύκολο, μπορείς να μεταφέρεις τα στοιχεία που μετράς σε αυτό το πεδίο. Το πιο δύσκολο είναι να μετρηθούν τα μέτρα της πολιτικής που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη και σχεδόν αδύνατο ε, να ε, αντιστοιχίσουμε τους δείκτες του αποτελέσματος, το outcome, το, το όμικρον από το SPO. Αυτό είναι δύσκολο λοιπόν για τους δικαιούχους, δηλαδή πιάνουν τόπο αυτά, φτάνουν στον τελικό δικαιούχο, τι νόημα έχουν όλα αυτά τα μέτρα, τι αποδίδουν και τι κέρδος έχουμε. Αυτό είναι το δύσκολο Επόμενη εμπειρία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, θα είμαι πιο σύντομος εδώ, Uh, Τι κάνει ο οργανισμός μας τώρα ε, για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στα πλαίσια του άρθρου 2 δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα να κοιτάμε ξεκομμένο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το ξεκομμένο και το ε, αυτόνομο που λειτουργεί σε ένα οδέτερο περιβάλλον είναι ευρύτερο παγκόσμιο το πλαίσιο. Λοιπόν, είτε θα στέλνουμε τα ευρωπαϊκά στοιχεία ε, σε διεθνές επίπεδο για να χρησιμοποιηθούν, παράδειγμα UPR, ή ε, θα εντοπίσουμε τον αποδέκτη. Δηλαδή, ας πούμε, σε οποιαδήποτε διεθνή ε, σύμβαση ε, έχουμε κάποια στοιχεία κομβικά, κεντρικά που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μην ξεχνάτε ότι το 2005, πριν από 10 χρόνια στη Βαρσοβία, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεταφέρει όλα τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ που τότε συμφωνήθηκαν ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Άρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το θέμα δεν είναι μόνο τα πρότυπα και οι προδιαγραφέ, αλλά είναι και οι φορεί που εφαρμόζουν όλα αυτά. Καλό είναι να μεταφέρονται σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε ε, ποιοι είναι οι φορείς αυτοί που τα ε, μεταφέρουν ε, οι διαμεσολαβητές, συνήγοροι του πολίτη, δικαστήρια αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή οτιδήποτε αποφασίζεται με αλφαγιώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεταφέρεται και οι φορείς που το διαχειρίζονται, οι αποδέκτες είναι όλοι αυτοί. Μπορεί αυτό να είναι υπομορφή συνεδρίου ή ετησίου διαλόγου στο Συμβούλιο, αλλά κάπως πρέπει να γίνει ε, μαζί με τους ενδιαφερομένους και τους δικαιούχους, αλλιώς χάνουμε την ε, υπόθεση αυτή. Και ε, κλείνω με μία πρόταση κάπως λειτουργική. Βεβαίως υπάρχουν ήδη πολλά στοιχεία και δεδομένα με τα διάφορα συστήματα ΟΗΕ, Συμβολίο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχουν και μετράνε διάφορα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχεις πρόσβαση. Ούτε οι εμπειρογνώμονες δεν γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο έχουμε περίπου 50 εκθέσεις παρακολούθησης και αναφορές για τα κράτη-μέλη σε διάφορα συστήματα και επίπεδα. Οπότε, ε, όχι, καταλαβαίνετε ότι αφού δεν μπορούν ούτε οι εμπειρογνώμονες να καταλάβουν τι τρέχει εκεί, φανταστείτε οι πολίτες θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούν όλα αυτά σε μια θηρίδα, one-stop shop ε, και το ιδεώδες θα ήταν online. Έχουμε το σύστημα ε, ε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ΕΦΙΣ. Εμείς πάντα μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, παρόλο που τώρα είμαστε στο άρθρο 2. Υπάρχει όμως ένας λόγος. Ο χάρτης θεμελιώδη δικαιωμάτων καλύπτει γύρω στο 80% των αρχών και αξιών του άρθρου 2 και αντανακλά τις αξίες του άρθρου 2 με πιο λεπτομερή τρόπο και ίσως και με πιο μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Σε συζητήσει για το άρθρο 2 λοιπόν έχουν τεράστια σημασία τα θεμελιώδη δικαιώματα και το να συσταθεί ένα σύστημα που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία θα δώσει και μεγαλύτερη προβολή σε κάποια διεθνή στάνταρ που ισχύουν όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να τα έχει αποφασίσει η ίδια. Ε, είναι ο ΙΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, επαναλαμβάνω. Και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εδώ επανέρχομαι στην εισαγωγή μου, συμφώνησαν επί δύο αρχών. Θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση για όλα τα κράτη-μέλη και αυτό θα πρέπει να γίνεται καλύτερα, μάλλον θα γίνεται με αντικειμενικούς και αξιόπιστους ε, αριθμούς και στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρνάτε Μαγκίνη, που, ε, μέλος της Επιτροπής της Βενετίας. Έχετε κάποια παρουσίαση? Θα εμφανιστεί η παρουσίαση σας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα. Δεν θα χρονοτριβήσω παρουσιάζοντας την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη γνωρίζετε. Είναι ανεξάρτητος συμβουλευτικός φορέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει 60 κράτη-μέλη που συμμετέχουν, πάνω από τα 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρα έχει επιρροή και εκτός της Ευρωπαϊκής Επίρου. Η Επιτροπή αυτή ε, της Βενετίας ασχολήθηκε με το κάτω δικαίου ποικιλοτρόπος Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Θέματα κράτους δικαίου εξετάσαμε, διάφορες χώρες, πάρα πολλές χώρες, ποικιλοτρόπως. Κάναμε λοιπόν αποτιμήσεις συνταγμάτων, νομοθετημάτων, κατόπιν αιτήματο συνήθως το κάνουμε αυτό. Εξετάσαμε θέματα κράτους δικαίου που ανεφάνισαν επίσης και συστημικά προβλήματα στον αφορά το δικαίου, πάντα κατόπιν αιτήματο του κράτους ή του φορέα που έχει δικαίωμα να ζητήσει γνωμοδότησή μας. Το 2011 εκπονήσαμε μια γενική έκθεση στον αφορά το δικαίου κατόπιν αιτήματο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και αυτή η έκθεση εξετάζει την έννοια του κράτους δικαίου, το κράτος δικαίου, το Rechtsstaat, το État de droit. Κατανοήσαμε βέβαια ότι είναι μεγάλο θέμα το δόγμα αυτό τι σημαίνει, τι καλύπτει ακριβώς. Ε, καταλάβαμε ότι είναι απίθανο να καταλήξουμε συμφωνία όσον αφορά τον, ορισμό του κράτους δικαίου παρόλο που υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που μας άρεσαν όπως αυτός του Τόμ Μπίγκαμ. Καταλάβαμε επίσης ότι ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο και το πολιτικό πλαίσιο υπήρχαν κάποια βασικά στοιχεία κοινά για όλους. Εδώ λοιπόν το 2012 κινηθήκαμε προς μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το κράτος δικαίου. Αντιληφθήκαμε ότι το κράτος δικαίου ίσως ήταν λιγότερο το αντικείμενο της προσοχής αυτό κάθε αυτό διότι είναι ένας από τους πυλώνες του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός εποπτείας. Αναφέρεται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφέρεται σε σχέση με ζητήματα δικαιοσύνης για δίκες, δίκες αλλά σπανίως αναφέρεται συστηματικά, με συστηματικό τρόπο, άρα είχε νόημα να παραχθεί ένα εργαλείο το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα για ορθή και συνεπή ερμηνεία της ενίας του κράτους δικαίου, ούτως ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή αυτού. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εστιαστούμε επί της εφαρμογής του κράτους δικαίου, αντί να συζητούμε εκτενώς την έννοια και ποια στοιχεία περιέχονται. Ξεκινήσαμε λοιπόν με, αυτό τον, αυτή τη λίστα των διαφόρων στοιχείων που έπρεπε, των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται. Είχαμε μια σύντομη, ένα σύντομο κατάλογο στην έκθεσή μας το 2011, συνεχίσαμε την επεξεργασία. Έχουμε τρία συστήμα, τρίες βαθμούς, πέντε συστήματα βαθμολόγησης που υποδιαιρούνται σε πέντε υποπαραμέτρους, νομιμότητα, δηλαδή η επικράτηση του νόμου, ασφάλεια δικαίου, απαγόρευση αυθερέτου προσεγγίσεως και κατάχρησης εξουσίας, ισότητα ενώπιον του νόμου, ε, μη διάκριση, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστικού κλάδου, δικαιοσύνη όσον αφορά την απόδοση δικαιοσύνης και συνταγματική δικαιοσύνη αν υπάρχει τέτοιο σύστημα σε μια χώρα. Λοιπόν, αυτές οι προδιαγραφές ε, συνοδεύονται από επεξηγηματικά σημειώματα ούτως ώστε να επεξηγούμε Έχουμε ένα ερωτηματολόγιο, λοιπόν, αυτό κατάλαβε ένα ερωτηματολόγιο. Ε, η βαθμολογία γίνεται εν είδη απαντήσεων σε ερωτήσει. Τα επεξηγηματικά σημειώματα εξηγούν τι εννοούμε και παραπέμπουν στι πηγέ. Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΔΕΚ ο, ή τα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε αποσαφηνίζουμε ακριβώ τι προσπαθούμε να εντοπίσουμε, τι εννοούμε με τι ερωτήσει. Και μετά έχουμε έναν κατάλογο συγκεκριμένων προδιαγραφών, προτύπων εκεί εξηγούμε από πού προέρχονται οι ερωτήσεις, ποια είναι η κοινή βάση, η ευρωπαϊκή και η διεθνής για, την, για τον σχηματισμό των ερωτήσεων. Λοιπόν, ε, έχουμε νομική βαθμολογία. Προσπαθούμε να, να καλύψουμε συνταγματική και νομική δομή, όπως αυτές οι δομές ερμηνεύονται στη συγκεκριμένη χώρα, ποια νομοθεσία ισχύει, ποια είναι η νομολογία των δικαστηρίων συγκεκριμένης ε, χώρας. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα, ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα, οι ερωτήσεις είναι διορίζονται επιμονή μου βάσος οι δικαστές ή μέχρι της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως. Αυτή είναι μια ερώτηση που απαιτεί εξέταση των κανόνων που ισχύουν στη χώρα, του συντάγματος αν υπάρχει συνταγματική βάση, του νόμου, των αρχών, της νομολογίας αν αυτή τυχόν υπάρχει. Άρα είναι νομική νομικό ερώτημα, νομική βαθμολόγηση εδώ. Τα περισσότερα αυτά συστήματα βαθμολόγηση είναι νομική φύσεω και κάποια αφορούν ε, την πραγματική κατάσταση ε, και εδώ συμπληρώνουμε τη νομική βαθμολογία. Ο κατάλογος αυτός με τις ερωτήσεις παραμένει νομικής φύσεως, άρα δεν μπαίνουμε σε άλλους τομείς. Λοιπόν, στην ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου, παραδείγματο χάρη, ερώτηση θεωρεί το κοινό ότι ο δικαστικός κλάδος είναι ανεξάρτητος. Το κοινό πώς αντιλαμβάνεται ενδεχόμενες πολιτικές επιρροές και χειραγωγή όσον αφορά τον διορισμό και την προαγωγή των δικαστών υπάρχουν ε, διορίζονται βάσει του συντάγματος για μια μόνιμη θητεία ε, ίσως όμως ο λαός να μην θεωρεί ότι επικρατεί διαφάνεια, ότι είναι ανεξάρτητος ο διορισμός και δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής χειραγώγησης. Και μετά με άλλες ερωτήσεις προσπαθούμε να εμβαθύνουμε την όλη ανάλυση. Προ, προφανώς για κάθε τέτοιο σύστημα βαθμολόγησης υπάρχουν και δυνατότητες πηγές επαλήθευσης. Τα κείμενα που ισχύουν για ένα νομικό κείμενο, νομικές αξιολογήσεις από την Επιτροπή Βενετίας, από, το, από τους ε, φορείς εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, από, άλλους, από άλλες πηγές. Λοιπόν, για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί και τη βαθμολόγηση. Έχουμε τους πολλαπλές πηγές, το ΣΕΠΕΖ, ε, υλικό από τους φορείς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, σφιγμομετρήσεις, υλικό από την κοινωνία των πολιτών, διάφορα άρθρα, ε, αυτές είναι διάφορες πηγές. Γιατί το κάναμε αυτό, ποια είναι η φύση αυτού του συστήματος βαθμολόγησης και ερωτήσεων. Ξεκινήσαμε στην Επιτροπή της Βενετίας δεχόμενοι ότι το κράτος δικαίου ε, είναι κάτι που συνεχώς ε, ανανεώνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Το να πετύχουμε το κράτος δικαίου να ολοκληρωθεί είναι θέμα πολυεπίπεδο και σταδιακής προσέγγισης. Κάθε χώρα προχωρά προς το κράτος δικαίου. Καμία χώρα δεν θα φτάσει πλήρως, είναι μια εφαπτώμενη πορεία. Κάποιες χώρες είναι πιο πριν, αλλά ε, συνέχεια υπάρχει πρόοδος προς τα εκεί. Οπότε έχουμε αυτό τον κατάλογο που περιέχει ερωτήσεις, αλλά δεν θέλουμε απλώς να συμπληρώνουμε διάφορα κουτιά και να λέμε αυτό είναι εντάξει, το άλλο είναι εντάξει. Δεν σημαίνει ότι αν όλες οι απαντήσεις δεν είναι θετικές ότι το κράτος δικαίου δεν ισχύει σε μια χώρα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, όλες οι χώρες έχουν ε, ισχυρά σημεία και αδυναμίες. Η προσέγγιση δεν είναι ή ε, άσπρο ή μαύρο. Η κυρία Μίχου λοιπόν ε, το ανέφερε επανειλημμένα. Η αξιολόγηση του κράτους δικαίου είναι περιπλακότατο εγχείρημα. Μία απάντηση σε μία ερώτηση. Παρόλο που υπάρχουν παράμετροι και βαθμοί και είναι απλουστευμένοι και η προσπάθεια είναι προσπάθεια απλούστευσης που βασίζεται σε κατάλογο ερωτήσεων, αλλά παρόλα αυτά οι απαντήσεις σε ε, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Πρέπει να τις επεξεργαστούμε όσο ενδείκνυται. Σφαιρικός πώς, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο αριθμούς, όχι μόνο αρνητικές ή καταφατικές απαντήσεις. Η αξιολόγηση λοιπόν του καταλόγου αυτού είναι ε, σφαιρική. Λαμβάνουμε υπόψη μεγάλο αριθμό στοιχείων, πηγών, ισροών πληροφοριών. Για ποιον προορίζεται αυτός ο κατάλογος. Για διάφορους φορείς. Η Επιτροπή της Βενετίας δεν παρήγαγε τον κατάλογο αυτό για συγκεκριμένο χρήστη. Θα χρησιμοποιηθεί από την Επιτροπή της Βενετίας βεβαίως όταν θα διενεργήσει αυτή μια αξιολόγηση ενός θέματος που αφορά το κράτος δικαίου θα βασιστεί σε αυτόν τον κατάλογο βαθμολόγησης. Όμως, ο κατάλογος αυτός αφορά και τους θεσμικούς φορείς, τα κοινοβούλια, τις αρχές κρατών που θα ήθελαν να προβούν σε μια αξιολόγηση του επίπεδου συμμορφώσεως με το κράτο δικαίου στη συγκεκριμένη χώρα, η κοινωνία των πολιτών που θα χρησιμοποιήσει τον κατάλογο και μας προσέγγισαν αρκετές μη κυβερνητικέ οργανώσεις πολλών χωρών που θα ήθελαν να έχουν κάποιο προσανατολισμό σχετικά με τη διάθρωση των αξιολογήσεών τους για το κράτος δικαίου σε μια χώρα και να το προσεγγίσουν το θέμα με καλύτερο τρόπο. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από διεθνείς οργανισμούς. Όταν ξεκινήσαμε την κατάτηση του καταλόγου, ο μηχανισμός αυτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν υφίστατο. Θεωρήσαμε όμως ότι θα μπορούσε να ταιριάξει στην όλη προσπάθεια. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα. Τι είναι το καινούριο για τον κατάλογο αυτό με τη βαθμολόγηση. Οι βαθμοί, οι πηγές ε, επαλήθευσης, οι μέθοδοι δεν είναι κάτι καινοφανές. Ο προλαλής σας ανέφερε ότι υπήρχαν πολλά στοιχεία διαθέσιμα οι φορεί εποπτείας του Συμβουλίου τη Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΦΡΑ, ε, ο ΙΕ, οι κοινωνίε των πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλέ πηγέ που χρησιμοποιούνται. Τα πάντα υπάρχουν. Αλλά αυτό που θεωρούσαμε ότι έλειπε ήταν μια σφαιρική προσέγγιση. διεξοδική ανάλυση των θεμάτων. Δεν είναι το ίδιο να εξετάζει κανείς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα χωρίς να εξετάζει το γενικότερο πλαίσιο. Και όταν το κάνουμε αυτό λοιπόν, τι κάνουμε. Πάντα ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση. Πάντα χρησιμοποιούμε την ε, το ίδιο σύστημα βαθμολόγησης. Είμαστε διαφανείς όσον αφορά τις πηγές μας. Οι χώρες όταν αξιολογούμε την ομοθεσία τους κατανοεί η χώρα σαφώς τι ακριβώς χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε συνεχώς για όλες τις χώρες πάντα ε, το ίδιο σύστημα βαθμολόγησης. Είμαστε αντικειμενικοί όσο πρέπει. Όσο μπορούμε, όσο υπήρξαμε με άλλες χώρες. Ποια είναι η κεντρική ιδέα. Να παράγουμε σαφείς κανόνες του παιχνιδιού. Όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, όταν εξετάζουμε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου σε μια χώρα, η χώρα αυτή πρέπει να γνωρίζει τι εννοούμε. Βάσει ποιου κινούμεθα, ποιο είναι το εγχείρημα. Και η χώρα θα πρέπει να γνωρίζει ότι έκαναμε ακριβώς το ίδιο σε κάθε περίπτωση όταν ασχοληθήκαμε με θέματα κράτους δικαίου. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Το πλαίσιο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις ενδεικνυόμενες συμβουλές από την Επιτροπή της Βενετίας, μπορεί να ζητήσει όπως έκανε κατά το παρελθόν ή να βασιστεί σε αξιολογήσεις και γνωμοδοτήσεις που έχουμε εκπονήσει για συγκεκριμένους νόμους χώρας, μπορεί να ζητήσει θεωρητικά πάντα να αξιολογηθεί το κράτος δικαίου επί τη βάση του συνολικού καταλόγου με το ερωτηματολόγιο ή μέρος αυτού. Προφανώς όμως ο κατάλογος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιονδήποτε το ζητά ε, απευθείας χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση της Επιτροπής της Βενετίας. Ε, επόμενη διαφάνεια. Θα κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι η πλήρης επίτευξη τη εφαρμογής του κράτους δικαίου είναι κάτι ουτοπικό, καμία χώρα το έχει πετύχει αυτό. Κάθε χώρα μπορεί καταρχήν θεωρητικά να το πετύχει. Η συμμόρφωση με το κράτος δικαίου θα πρέπει συνεχώς να ελέγχεται και ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός ούτε τελικός. Το checklist όπως το λέμε θα εισιτηθεί κανονικά τον Μάρτιο. Συνεχώς θα εξελίσσεται, παρόλα αυτά το χρησιμοποιούμε και ελπίζουμε ότι θα παραγαγεί τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις. Έχουμε τον τελικό ομιλητή. Δόκτωρ Τζερίντα Μπεωράλ από το Κέντρο για το Κράτος Δικαίου του Μπίνγκαμ από το Βρετανικό Ινστιτούτο του Διεθνούς και Συγκριτικού Νόμου, η κυρία Τζελίντα και θα αναφερθεί σε δείκτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παγκόσμιους δείκτες και θα δώσει κάποια θέματα όσον αφορά τον εντοπισμό εθνικών δικτών ε, ουσιαστικά από τη Γερμανία και το Ενωμένο ε, Βασίλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια άλλη ε, διάσταση που θα διαμορφωθεί τα επόμενα 15 χρόνια σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στο πλαίσιο των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων που συμφωνήθηκαν στη Νέα Υέρκη από τη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο του 2015. Βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις βασικές ενότητες της παρουσίασής μου. Μία σύντομη παρουσίαση του σε τι διαφέρουν οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι από τους προηγούμενους ε, αναπτυξιακούς ε, στόχους της χιλιετίας και, τον, και τους ε, στόχους του 16 για το κράτος δικαίου. Ποια είναι, η διαδικασία σήμερα για την οδοποιησμό καθολικών δικτών και τέλος να συζητήσουμε δύο παραδείγματα εθνικών διαδικασιών στον Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. MDGs και SDGs της χιλιετίας, αναπτυξιακή στόχη και βιώσιμη αναπτυξιακή στόχη. 2015 με 2030 οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι. Είναι λοιπόν ολιστική η κατανόηση των ε, βιώσιμων στόχων. Έχουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Και για πρώτη φορά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται και οι απόψει τη κοινωνία των πολιτών. Έγιναν διαβουλεύσεις οι οποίες και ενσωματώθηκαν στα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, είναι καθολικοί στο πεδίο εφαρμογή τους. Δεν αναφέρονται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά σε όλα τα κρατημέλη του ΟΗΕ. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα τον 16ο στόχο. που αφορά το κράτος και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεσμεύει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα συστήματά τους ως προς αυτές τις δύο διαστάσεις. Αυτό αναφέρεται όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες. Και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία λοιπόν, για παράδειγμα, μπορούν να βελτιώσουν το σύστημα κράτους δικαίου. Ένα άλλο καινοτομικό στοιχείο των ε, βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και θα ήθελα να επικεντρωθώ ιδιαίτερα στον 16ο στόχο που έχει και περιλαμβάνει ακριβώς την πτυχή της πρόθεσης του κρατου δικαίου σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο και η συμπρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Ο απόδραστος αυτός σκοπός ε, διαμορφώνονται και από πιο συγκεκριμένους στόχους. 16-3 συγκεκριμένα Βλέπουμε τον στόχο 16.3 που δεσμεύει τα κράτη-μέλη να προωθούν το κράτος δικαίου σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλίσει ίση πρόσβαση για όλους. Και άρα εδώ πέρα προσέχουμε ότι μιλάμε για προώθηση, όχι εξασφάλιση κράτους δικαίου. Είναι μια διαρκής διαδικασία και εξασφάλιση της πρόσβησης στη δικαιοσύνη. This is the target and, um... Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρούμε και τους σχετικούς δείκτες για το πώς μπορεί να προσμετρηθεί ο στόχος αυτός ανακράτος μέλος. Στα αριστερά λοιπόν βλέπετε στη διαφάνεια μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, στατιστικολόγων, που έχει εντοπίσει τους δείκτες για τους ε, εκάστοτε στόχους, συμπεριλαμβανομένου και του 16.3. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα γράμματα. Είναι με βασίλειο λοιπόν Προεδρία, Τανζανία, Ουγγάντα, Μποτσουάνα, Καμερούν, Πράσινο Κροτήρι, Σενεγάλη, Αλγερία και στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Καναδάς, Γαλλία, Αμερική, ε, κάτω Σουηδία. Μιλάμε λοιπόν για ένα σώμα τεχνικών, στατιστικολόγων. Εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι μάλλον από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των χώρων αυτών. Οι οποίοι και υπέβαλαν μία σειρά προτάσεων. Τρεις εξ αυτών σας παρουσιάζω λοιπόν εδώ. Αντίστροφα, οι πρώτοι δύο περιλαμβάνονται στο σχέδιο κειμένου, το οποίο και θα παρουσιαστεί στην ε, Στατιστική Υπηρεσία του ΟΗΕ το Μάρτιο του 2016 και μετά θα συζητηθεί σε πολιτικό σώμα του ΟΗΕ. Θα παρουσιαστεί λοιπόν στους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Δυστυχώς η τάση είναι να αποδυναμώνονται οι δείκτες αυτοί. Βλέπετε λοιπόν από τους πρώτους δύο δείκτες ότι εστιάζονται κυρίως στην ποινική δικαιοσύνη. Δεν καλύπτουν δηλαδή τον πυρήνα του στόχου 16.3. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ποινική, δικονομική δικαιοσύνης. Είναι πολύ στενή λοιπόν οι δείκτες αυτοί ο τρίτος, ήταν, ε, ο δείκτης είναι ο πρώτος που προτάθηκε και εξακολουθεί να υποστηρίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και από τις μεγάλες ε, παγκόσμιες οργανώσεις, την Παγκόσμια Τράπεζα, το UNDP κτλ. Πρόκειται για έναν πιο ευρύ δείκτη για να προσμετράτε η αναλογικότητα, μάλλον το ποσοστό εκείνων που έχουν ζήσει διένεξη τα τελευταία, τους τελευταίους 12 μήνες και που είχαν πρόσβαση σε δικαίη, επίσημη, ανεπίσημη, εναλλακτική και παραδοσιακή μορφή αντιμετώπισης μηχανισμού διενέξεων. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο τη θεσμική διάσταση, αλλά και την αντίληψη του κόσμου, γιατί μιλάμε για δίκαιη τέτοια μορφή επίλυσης διαφορών. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά τα συλλέγουμε με συγκεκριμένες μελέτες. Και στόχος λοιπόν ήταν να συμπεριληφθούν μελέτες στα νοικοκυριά, άλλος ένας ε, άλλη μια κατηγορία που θα μπορούσε να μας δώσει τέτοιου είδους πληροφορίες. Για να αποκτήσουμε τέτοια στοιχεία, τα οποία δεν έχουμε στη διάθεσή μας στην παρούσα φάση. Εν συντομία τώρα, να σας παρουσιάσω και τα δύο παραδείγματα. Πέρα από τους παγκόσμιους ε, δείκτες, σε επίπεδο κράτους και σε περιφερειακό επίπεδο, οι εθνικοί και περιφερειακοί δείκτες μπορούν να εφαρμόσονται στα εκάστοτε επίπεδα. Η διαδικασία για τον εντοπισμό των δικτύων αυτών είναι διαφορετική, καθότι κάθε κράτος έχει διαφορετικές αρχές. Ένα καλό μοντέλο είναι το γερμανικό γιατί είναι και το πιο προηγμένο. Πέρα από τον εντοπισμό προτεραιοτήτων και των τομέων προτεραιότητας, περιλαμβάνει και δύο επίπεδα ελέγχου. Το πρώτο είναι το κρατικό συμβουλευτικό συμβούλιο, που περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες, που εξετάζουν τις πολιτικές προς την κατεύθυνση επίτευξης και υλοποίησης των στόχων και μια κοινοβουλευτική επιτροπή συναποτελούμενη από όλα τα κόμματα που εκτιμά την επιτυχία και την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων. Για το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε περιφέρεια έχει λάβει αυτόνομα μέτρα. Η Ουαλία και η Σκοτία στην παρούσα φάση έχουν ξεκινήσει η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Στην Αγγλία δεν έχουν λεφθεί ε, μέτρα ακόμη. Ενδεχομένως να υπάρξει όμως κάποια πιο κεντρική δράση σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε 20-25 λεπτά περίπου για ερωτήσεις. Ας πάμε λοιπόν κατευθείαν στους κοιόδης. Να ακούσουμε τον κύριο Έγγελ. Στα αγγλικά ο κύριος Έγγελ. Έχω μια γενική ερώτηση προς όλους. Που δεν είναι και τόσο ερώτηση. Το οποίο προσωπικά έχω εξαγάγει από όλες προσπάθειες να καταλάβω τι μου γίνεται εδώ. το να καθορίσουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κράτος δικαίου ή τα κράτη είναι σαν να λες για να δούμε αν η Κίνα είναι ελεύθερη οικονομία. Έχουμε πέντε πρότυπα, ο καθένας κάνει τα δικά του, Αμερική, Αυστραλία κτλ. Κάποια στιγμή θα καταλήξουμε ε, ότι είναι κράτος δικαίου, όχι επειδή είναι, αλλά επειδή εκεί πρέπει να καταλήξουμε. Αυτό ισχύει και για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι, στα πρότυπα και τις προσδιαγραφές τους, ξέρω ότι έχει στάνταρ, αλλά θα μπορούσα εύκολα να ε, αναφέρω 5-6 ε, μέλη, ε, κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου πιστεύω ότι αυτές οι προδιαγραφές για το κράτος δικαίου, δημοκρατία και κάτι άλλα απέχουν μίλια από ένα κράτος δικαίου πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τραβήξει κανένα αυτή το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και καιρό και θα έχει τους λόγους του μάλλον. Λοιπόν, Ακούγοντας εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες όπως εσείς, ε, πού καταλήγω ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν είναι λογιστική. Κατά την άποψή μου, Μπορεί να υπάρχουν εργαλειοθήκες, δείκτες, φόρμουλες και δεν ξέρω τι άλλο, κορσέδες, για να μπορέσει κανείς να μελετήσει ότι κάτι λειτουργεί και κάτι όχι. Ιδιαίτερα στην Ήπειρό μας, όπου έχουμε τεράστιες διαφορές στη διακυβέρνηση. Έχουμε ζήσει και χούντες, ορισμένοι πιο πρόσφατα, άλλοι πιο παλιά. Έχουμε κράτη που έχουν ε, παράδοση χιλιετιών κράτους δικαίου και διακυβέρνησης, χωρίς να έχουν καν γραπτό σύνταγμα ε, και μπορεί ο Πρόεδρος να θυμάται ποια χώρα εννοώ. Και άλλες χώρες που έχουν αυτή την παλιά παράδοση. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση της κυρίας ε, Γρανάτα Μενγκίνη που είπε όταν η Επιτροπή Βενετίας θεώρησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη ορισμών σε αυτά γιατί χρειαζόμαστε συνένεση για κάποια βασικά στοιχεία και θεμελιώδη. Αυτό θέλω και εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επανέρχομαι σε κάτι που γνωρίζει η Σόφη Ινετφέλτ και κάποιοι άλλοι, γιατί είμαστε σκιώδεις ηγητές. Είναι να δούμε αν υπάρχει ε, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης, μια ευρωπαϊκή λογική. Έχουμε αποφασίσει με ποιο τρόπο θέλουμε να διοικούμεθα, να μας κυβερνάνε. Μπορεί να είναι τα στοιχεία αυτά και μετρήσιμα και ε, ποσοτικά, αλλά κυρίως είναι χειροπιαστά και ε, ε, αισθανόμαστε. Δηλαδή, να μην αυθαιρετεί το κράτος, να μην υπάρχει διαφθορά, να προβλέπεις τι θα κάνει το κράτος. Να υπάρχει μια προβλεψιμότητα και να καταλαβαίνει ο πολίτης και να αισθάνεται ότι ξέρει τι του γίνεται ότι το κράτος και η κοινωνία, η συντεταγμένη κοινωνία κάνει αυτό που πρέπει και αν δεν το κάνει μπορούν να την αλλάξουν τη διοίκηση. Ε, κάπως έτσι νομίζω θα πρέπει να κινηθούμε και να εστιάσουμε. Δεν με πειράζουν και οι πίνακες επιδόσεων και οι δείκτες και όλα αυτά που μετράμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι πιο πολύ για τα τεχνικά δεν μετράνε πράγματα τόσο εθέρια όπως είναι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η κυρία Μόνικα Μπένοβα. Mm. E, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, πολύ καλή ε, η σημερινή ακρόαση και πάρα πολύ επίκαιρη και εύστοχη. Έχουμε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας στην Επιτροπή μας ε, και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτή τη βδομάδα είχαμε εδώ δημοσιογράφους από τα κράτη-μέλη σε ένα σεμινάριο για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Εχθές συναντήθηκα επί δύο ώρες με δημοσιογράφους από τη Σλοβακία και μου έκαναν ερωτήσεις για τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε σε σχέση με ε, τη μη τήρηση κάποιων υποχρεώσεων ε, από τα κράτη-μέλη. Με ρώτησαν δηλαδή τι θα γίνει αν ένα κράτος μέλος δεν, ε, υλοποιείται δεν υλοποιεί όσα έχει υποσχεθεί για τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες, ας πούμε. Ποιος μπορεί να μας αναγκάσει να τα εφαρμόσουμε για τη μετανάστευση τώρα. Ποιος μπορεί να αναγκάσει τη Σλοβακία να ε, υλοποιήσει όλα αυτά. Μεταξύ άλλων κρατών, η χώρα μου δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι πρόθυμη να συμμετέχει σε κοινέ αποφάσεις ε, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στα κράτη-μέλη δημιουργούνται καταστάσεις που αγγίζουν τα όρια και τα εξαντλούν πολλές φορές της νομιμότητας και του κράτους δικαίου. Και τώρα ε, υποστηρίζονται όλα αυτά και νομοθετικά από νέους νόμους που περνάνε από κοινοβούλια. Εσείς πώς το βλέπετε και πώς το βλέπουν και οι οργανισμοί τους οποίους εκπροσωπείτε εδώ. Για τα κράτη-μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι δίστροπα ας πούμε ή απίθαρχα. Πώς ε, θα ε, επιβάλλονται κυρώσεις. Στη δική μας Επιτροπή συζητάμε συχνά για τη μη τήρηση θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Και οι περισσότεροι από εμά τα γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, είμαστε σκιώδεις ηγητές συχνά και ασχολούμαστε πολύ και για μεγάλο διάστημα με την ε, τήρηση, των, την εφαρμογή των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη για το σεβασμό τους. Έχουμε εγκρίνει και πολύ ωραίες εκθέσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν κατονομάζουμε κανέναν, δεν φύγουμε κανέναν, ε, αλλά κάπου πρέπει να δείχνουμε και κάποια συνέπεια. αν δεν χρησιμοποιούμε το σύστημα κυρώσεων που προβλέπεται, αν δεν τηρούμε εμεί τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα, τι θα γίνει. Θα παραμείνουμε μια λέσχη συζητήσεων που μπορεί να κατονομάζει τα προβλήματα, αλλά μέχρι εκεί δεν προχωρήσει συγκεκριμένες λύσεις για τους πολίτες. Και έχουμε σήμερα μια τέτοια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μιλούν για το θάνατο της Σέγγεν, για διάφορους κανόνες καινούριου. Εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε εμείς. Και να δούμε τι κάνουμε με τα ίδια μας τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται. Πρέπει να υπάρχει σύστημα βολής κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Καρκόπ, πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Με όλους αυτούς τους κανόνες, εποπτεία, συστήματα βαθμολόγησης κλπ. Όλα αυτά καλά και άγια. Πρέπει να δούμε όμως πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά. Υπάρχει αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ κυριαρχίας κρατών μελών με την εφαρμογή του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πολλές κουβέντες γίνονται κυρίως σε αυτή την Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο. Τακτικά κουβεντιάζουμε κάποιες χώρες. Κατά πόσο θεωρούμε ότι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε εντελώς αντικειμενικοί σε ένα πολιτικό σύστημα δύσκολο να κρίνουμε αντικειμενικά και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε όσα συστήματα βαθμολόγησης θέλετε. Αλλά στο κάτω-κάτω πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά από αυτό. Τι εξουσίες έχουμε. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά. Καλό να μιλάμε για ακυρώσεις. Αλλά και αυτό γίνεται θέμα για υποκειμενική συζήτηση. Επανειλημμένα έχει γίνει στην Επιτροπή. Επικοδομητική συζήτηση, άκρως ενδιαφέρουσα, αλλά υπάρχει αυτή η βασική σύγκρουση που ανέφερα. Και όσο συνεχίζεται αυτή, και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί όπως απαιτείται, πολύ δύσκολο να βρούμε κάποια διέξοδο. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπινέλη, η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέση και ερωτήσεις. Η κυρία Γκρανάτα Μεγκίνη μας είπε κάτι. Ότι η πλήρης επίτευξη του κράτους δικαίου είναι κάτι ουτοπικό. Το να λέει κανείς κάτι τέτοιο ελαφρά την καρδία είναι επικίνδυνο. Είναι δύσκολη η πλήρης επίτευξη του κράτου δικαίου, αλλά δεν είναι κάτι τοπικό, διότι το τοπικό είναι κάτι ανύπαρκτο. Είναι σαν να λέμε ότι είναι τοπικό το να θέλουμε, η μεταρρύθμιση είναι κάτι α, οτοπικό. Άρα η, δια, η συντήρηση είναι το μόνο που μένει. Δεν έχουμε επανάσταση, δεν έχουμε μεταρρύθμιση πια. Άρα δεν μένει τίποτα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού. Έχουμε διάχυτη παραβίαση των δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες, την ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη, που κίνδυνος να λέμε, είναι επικίνδυνο να λέμε το κάτω δικαίου είναι ουτοπικό. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές συζητήσεων για το κάτω δικαίου. Το κάτω δικαίου πρέπει να εφαρμόζεται. Δύο ερωτήσεις. Πρώτο από προς την κυρία Μίχου για το νέο σύστημα εποπτείας, για το εξάμεινο, είπατε ότι θα ελέγχεται κυρίως η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και πώς εφαρμόζεται αυτή στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να ρωτήσω, επ' αυτού υπάρχουν πολλές μελέτες για πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων του άρθρου 2 ή της χάρτας και των πολιτικών που αποφασίζονται το εξάμεινο. Οι μελέτες αυτές για παραβιάσεις άλλων δικαιωμάτων θα λαμβάνονται υπόψη στο εξάμεινο. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας για την αυτοεξαίρεση, για το opt-out που ζήτησε το Ηνωμένο Βασίλειο από το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Σύστημα και από τα δύο δικαστήρια. Αυτό μελετάτε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Έχω άλλα τρία μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα κλείσω τον κατάλογο. Όλοι έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα θέματα, σχετικά των θεμάτων. Παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη να είστε σύντομοι. Δύο λεπτά ο καθένας ο κ. Λόπες Αγγελάρ, Άννα Γκόμες και Σοφή. Χουάν Φερνάντο. Σε παρακαλώ δύο λεπτά. Ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία να ακούσω από τους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής ε, της Βενετίας και του Εβεράη για τον Οργανισμό θέμελι των Δικαιωμάτων, τι γίνεται με τους έντοντες ε, άσυλο στα κράτη-μέλη και ε, τι γίνεται και από πλευρά των κρατών μελών. Υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις, διαφορές στο πώς ε, σεβόμαστε και σέβονται τα κράτη-μέλη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά και για τους Αλλοδαπού ιδιαίτερα τι γίνεται με την περίπτωση της Ουγγαρίας, της Ισπανίας στα ανατολικά, στα νότια σύνορα, σε ό,τι αφορά τις ε, ε, επιστροφές ε, ετούντων άσυλο. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Γκόμες. Και εγώ χαίρομαι που έχουμε έχουμε μεθόδους και πρότυπα και ούτω καθεξής. Αλλά ας τα εφαρμόσουμε κιόλα να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση φρικτή. Με όρους ε, σχετικούς μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτά που πετύχαμε. Αλλά είναι λυπηρό, είναι λυπηρό να δούμε τι έχει συμβεί πρόσφατα και το πώς ε, δεν έχουμε ανταπεξέλθει δεν έχουμε έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το κράτος δικαίου ως μια ουτοπία. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα μας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη. Αν είναι τοπικό και δεν μπορούμε να το πετύχουμε έτσι κι αλλιώ. γιατί να το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχο σα και ο σωστό τρόπο παρουσίασης της κατάσταση. Εγώ Πραγματικά αξιολογώ τα πράγματα με πολύ λύπηρο τρόπο. Εγώ είμαι από μια χώρα τρόικας, όπου η τρόικα σήμαινε πιο πολύ φτώχεια, πιο, ανισότητα, μεγάλη ανισότητα, ένα τρίτο των παιδιών μας σε καθεστώς φτώχειας. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Και φυσικά διαφθορά, ανισότητα στα φορολογικά και όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απογοήτευσε και φυσικά αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Πού την καταπολεμάει η διαφθορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι να την κάνω την έκθεση αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε δράση, ενέργεια για κρίσιμες περιστάσεις και περιπτώσεις. Περιπτώσεις που είχαμε στη χώρα μου, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία. Τι κάνουμε. Όχι μόνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, με τη συμπεριφορά της Ουγγαρίας και τη συμπεριφορά της στην πρόσφατη κρίση των μεταναστών. Ακόμα και ο πρόεδρος Τάσκα ζήτησε πρόσφατα. Τους ζήτησε να α, ε, κρατούνται οι μετανάστες. Και τελευταία ερώτηση. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, πώς γίνεται να αγνοούν στόχοθετημένες ε, δολοφονίες ε, πολιτών της Ένωσης από ένα κράτος μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, ναι, ναι, διακόπτει ο Πρόεδρος, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Η κυρία Ιντφέλτ, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της σημερινής μα ακρόαση, γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία ακολουθεί ο κάθε συνάδελφο ενδεχομένω. Σα παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρο, δεν έχει ολοκληρωθεί η ακρόαση. Σα παρακαλώ, ησυχία. Δεν έχω το σφυράκι. Σας παρακαλώ, ησυχία. Θα συνεχίσω, λέει η κυρία Ιντσφέλτ. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση να κάνω. Και νομίζω καλό θα ήταν ε, αν το πάνελ θα μπορούσε να απαντήσει κυρίως τα ερωτήματα και τις ε, παρατηρήσεις για τους δείκτες. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Άκουσα τον κύριο Έγγελ και τον κύριο Κέρκοπ που εκφράζουν έναν κάποιον σκεπτικιστισμό για την ε, ανάπτυξη και εφαρμογή των δικτών. Να γνωρίζω ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι απλό και εύκολο. Το γεγονός όμως ότι είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό ή εντελώς αδυνατό να αναπτυχθούν δίκτες ή δείκτες. Δεν είναι μεζούρες, είναι δείκτες. Αυτή είναι η λειτουργία τους και νομίζω ότι μπορούν να προσμετρήσουν κάτι πραγματικό και απτό. Μία ερώτηση να κάνω προς τον κύριο ο οποίος μας μίλησε για προσπάθειες. Για το ΕΦΡΙΣ. Γιατί είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα τέτοιο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αν θα θέλετε να μας απαντήσετε και σας ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε χρόνο αρκετό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μίχου. Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ στις απαντήσεις που θα δώσει το πάνελ. Εκτός του πάνελ μπορούμε να συζητήσουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά όχι τώρα. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη Σοφή Συμφωνώ με το πρώτο που είπε, το κάτω δικαίου είναι σημαντικότατο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακολουθούμε αυτή τη στάση. Κάνουμε πολλές προσπάθειες για να ε, τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πολλές φορές οι προκλήσεις εμφανίζονται πιο γρήγορα από τις απαντήσεις που δίνουμε. Αλλά απαντούμε σε πολλές περιπτώσεις και συμμόρφωση και εφαρμογή και παραβιάσεις και για θέματα μετανάστευσης όλα αυτά τα θέματα αξιολογούνται. Για κάποια από τα θέματα που παρουσιάστηκαν από τα μέλη του πάνελ θέλω να πω το εξή. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εναλλακτικοί μηχανισμοί διευθετήσεως διαφορών ρυθμίζονται από δείκτε. σω χρειάζεται περαιτέρω κατάρτιση. Υπάρχουν στο σύστημα βαθμολόγηση, στο scoreboard που έχουμε, το πίνακα βαθμολόγηση. Και είναι συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρκεια τη τριετία που είχαμε το σύστημα αυτό. Τι θέλω να πω τελικά. Πιστεύουμε όλοι το κράτο δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό για το κάτω δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Ας εργαστούμε. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας. Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μακριά πάνω σε απτά ζητήματα. Ένας τομέα όπου χρειάζεται πρακτική προσέγγιση, πρακτική δουλειά. Οι δείκτε είναι κάτι πρακτικό. Και είναι η βάση επί της οποίας Εκτιμούμε την ε, υλοποίηση του κάτω δικαίου. Πρέπει να αποχωρήσω τώρα γιατί έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας. Εκτιμούμε την υπομονή σας που μείνατε εδώ. Ο κ. Στόγκενμπεργκ λοιπόν έχει το λόγο. Σύντομα παρακαλώ. Να απαντήσουμε και μπορεί να απαντήσετε και γραπτός. Δύο πράγματα. Συγκεκριμένη ερώτηση για το ΕΦΡΙΣ. Δεν έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για το σύστημα πληροφόρησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, γιατί σύμφωνα με την εμπειρία μας ε, ε, οι τράπεζες δεδομένων πρέπει να είναι βιώσιμες και θα πρέπει όλοι οι φορείς να συμμετέχουν και το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά καλό θα ήταν να δούμε τι κάνουν και άλλοι θεσμοί και να καταλάβουν ότι εδώ πρόκειται για κάτι το υποστηρικτικό. Για του δείκτες βλέπω ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα ότι οι δείκτες είναι για, για κάποιους ε, υπερβολικούς εμπειρογνώμονες και το θέμα δεν είναι οι δείκτες για τους δείκτες, ε, για τον έλεγχο, αλλά για την εφαρμογή, για την υλοποίηση. Και στο Συμβούλιο, ε, στην ετήσια συζήτηση για το κρατός δικαίου, θα μπορούσε να μπει αυτή η συζήτηση ότι για την υλοποίηση χρησιμεύουν οι δείκτε. Διότι η ισότητα σημαίνει ότι έχει και διαρθρωμένο διάλογο και για να διαρθρώσει ένα διάλογο χρειάζεσαι δείκτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ και πάλι. Σιμώνα, δύο προτάσεις να πεις. Κάτι λέει κυρία Νετφέλτ εκτός μικροφώνου. Ναι, θέλω και απαντήσει όμω να ε, ακούσω. Καταληκτικά και αλλιώ γραπτό τα υπόλοιπα. Έχουμε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία, καταξέρισε. Ευχαριστώ. Συντομότατα. Οι αξιολογήσει είναι απαραίτητες. Διενεργούνται από διάφορους φορείς. Υπάρχουν διάφορα θέματα που αφορούν τις κυρώσεις. Η αξιολόγηση είναι κάτι που προηγείται. Δεν έχει απαραίτητα το στόχο την επιβολή κυρώσεων. Ίσως έχει στόχο βελτίωση της καταστάσεως με διαφορετικούς τρόπους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διενέργεια των αξιολογήσεων βάσει αντικειμενικών, συνεπών και ισοτήμων κριτηρίων είναι κάτι που βοηθάει γενικά την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ, πολύ επικοδομητικό. Δόκτωρ Μπεκεράτς παρομοίως σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη, πολύ σύντομα. Η ιδέα του να έχουμε προσμετρήσιμους δείκτες είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για να πάμε κατά των επικρίσεων. Δηλαδή ότι το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη είναι έννοιες που δεν μπορούν να μετρηθούν. Και ότι είναι αποκλειστικά πολιτικές δεσμεύσεις και εξαρτώνται πολύ από την πολιτική βούληση και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος για την εφαρμογή αυτών. Εκτός αν έχουμε το πυρηνικό όπλο, όπως ανέφερα, ε, δηλαδή επιβολή κυρώσεων αν δεν εφαρμόστε κλπ. Είναι σημαντική οι δείκτες. Ευχαριστώ τους ομιλητές για την παρουσία τους, ευχαριστώ τα μέλη, διότι ήταν έξοχη η ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοθεί συνέχεια, ευχαριστώ τους κοιόδης και τα μέλη. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε να επενθυμίσω ότι ξεκινήσαμε την ακρόαση χωρίς να ξεκινήσουμε επίσημα τις εργασίες. Θα ξεκινήσω με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να κάνετε λίγη ησυχία, να καθίσετε. Έγκριση ημερησίας διατάξεως, αν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη. Να πω κάποια πράγματα πριν πάμε στην ψηφοφορία. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Γλωσσικό συνδυασμό, διερμηνία στα νέζικα, λετωνικά, ε, κροατικά και γολεδικά δεν θα είναι διαθέσιμα σήμερα. Λοιπόν, ε, έχουμε καθορίσει τους εισηγητές θα είμαι συγητή για την εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου για την, την εκκίνηση αυτόματης ανταλλαγής ε, στοιχείων για την καταχώρηση οχημάτων στην Λετωνία. Θα αναλάβω κατ' εξαίρεση αυτή την έκθεση. Η κυρία Βαλέρο Μποντέλ των Πρασίνων είναι συγγήτρια για την γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου για τον έλεγχο της απόκτησης και κατοχής όπλων. Αυτό είναι έτοιμα δυνάμει το άρθρο 54 ε, με την Επιτροπή ΙΜΚΟ και τελικά όσον αφορά τον καθορισμό εισηγητών σαν αποτέλεσμα συστάσεων των συντονιστών Έχουμε την κυρία Λάουρα Αγκαία τη CFTD, η οποία είναι εισηγήτρια για την γνωμοδότηση όσον αφορά την προετοιμασία της ε, μετεκλογικής αναθεωρήσεως του ε, πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και ποια είναι η πρόταση του Κοινοβουλίου πριν από την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, εγκρίνεται τις προτάσεις των συντονιστών. Μάλιστα, τις εγκρίνεται. Συνάδελφοι, λοιπόν, ερχόμαστε στην ψηφοφορία. Καταρχάς, να ελέγξω ότι όλοι έχετε τις ε, κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν κάποιος δεν έχει την κάρτα του, παρακαλώ να μας το επισημάνετε. Κανείς ε, δεν υπάρχει χωρίς την κάρτα του. Άρα δεν θα λάβουμε υπόψη ψήφο κάποιου που μετά θα πει κάτι διαφορετικό. Όλοι λοιπόν θα ληφθούν υπόψη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ονομαστική ψηφοφορία. Το λέω αυτό για τεχνικούς λόγους. Πολύ ησυχία βλέπω. <laughs> Περίεργο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Είναι σημαντική η ψηφοφορία που μας περιμένει. Ωραία. Επόμενο σημείο της διάταξης. Α, for balance, is there anyone late from any other group that could... Uh... Υπάρχει κάποιο που έχει καθυστερήσει από άλλε ομάδε. Λοιπόν, συνάδελφοι, επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ψηφίζουμε το συμπεφωνημένο κείμενο. Το συμφωνήσαμε στι διοργανικέ συζητήσει για την οδηγία για το ευρωπαϊκό PNR. Ο εισηγητή, ο κ. Κέρκοπ, θέλει να πάρει το λόγο. Καλώ. Έχετε δυνατότητα να πείτε κάτι μετά την ψηφοφορία. Εν τη αυτή περίπτωση, αν έχετε ε, την καλοσύνη να δεχτεί να το κάνει αυτό ο κ. Κέρκοπ. Λοιπόν, για την πρόταση οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την χρήση του ονόματο, επιβατών και στοιχείων για την πρόληψη εντοπισμό έρευνα και δίωξη ε, τρομοκρατικών αδικημάτων και σοβαρών εγκλημάτων. Εισηγητής είναι ο κ. Κέρκοπ. Ψηφίζουμε το συμπεφωνημένο κείμενο. Αυτό ήταν αποτέλεσμα διοργανικών συζητήσεων και ψηφίζουμε ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ αν έχετε ψηφίσει όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο εισηγητής θέλει να πει κάτι. Πρόεδρε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, θέλω να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους ε, εργαζομένους αυτή την Επιτροπή και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής ανεξαρτήτως των απόψεών τους. Ήταν μακρά διαδικασία. Χαίρομαι όλες ιδιαίτερως με το αποτέλεσμα τώρα που βγήκε στην Επιτροπή και αυτό δείχνει η δουλειά έχει γίνει και νομίζω είναι πολύ λογική απόφαση και είμαι ευγνώμων προς όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους που κατέβαλαν την προσπάθεια. Έληξη ψηφοφορία και συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Um, Συνάδελφοι, πάμε στα υπόλοιπα σημεία της ημερησίας διάταξης. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αποχωρήσετε ησύχως. Παρακαλώ όμως να αναχωρήσετε ησύχως, διότι πρέπει να πάμε στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ, αποχωρήστε με ησυχία. Επόμενο σημείο, σημείο 5, διαφάνεια, έλεγχος αικαιρεώτη Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η της γνωμοδότηση, η κυρία Γκυόμ. Τη συζήτηση του σχεδίου γνωμοδότηση λαμβάνει η χώρα. Πιο πολύ φασαρία βλέπω, παρά ησυχία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις εργασίες. Είχε διοργανωθεί η κοινή ακρόαση τον περασμένο μάτι με τις επιτροπές Τζούρι, Λίμπε, Αύκο και Κοντ προς μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου, διαφάνειας και κυριότητας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης ήταν τίτλος. Βασίστηκε εκρόαση σε μια έκθεση όσον αφορά το σύστημα κυριότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσης που συνετάχθη από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, Transparency International. Σαν συνέχεια που δίδεται στην ακρόαση, η Επιτροπή ΑΦΚΟ επεξεργάζεται μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η κυρία Γκυγιόμ, η συγγήτρια για την γνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ στην έκθεση πρωτοβουλίας θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς της. Εσύ έχει το λόγο και θα προσπαθήσω να κάνω συναδέλφους να είναι ήσυχοι. Σε έχει το λόγο. Σιλβί, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τι ε, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποια αναταραχή μετά την ψηφοφορία αυτή. Πριν το ξεχάσω, θέλω κάτι να διευκρινίσω για προθεσμίες. Ε, ε, que le dépôt des Anatolia. Yes, ψηφοφορία, ε, μάλλον οι τροπολογίες ε, μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου το μεσημέρι για να ψηφίσουμε στις 25 του ε, Γενάρη. Αρχίζω από το χρονοδιάγραμμα για να το ξέρουμε αυτό. Για το ίδιο το σχέδιο γνωμοδότησης θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για τη διαφάνεια και τα λέμε κιόλας. Ε, πολλές ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές γνωμοδοτούν για την έκθεση του συναδέλφου Γκίγκολτ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ίντα, Γιούρι, Ένβη και Κόντ εκτός από τη δική μας Επιτροπή γνωμοδοτούν. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τόσο πολλές γνωμοδοτήσεις, εγώ επικεντρώθηκα κυρίως σε θέματα που είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητάς μας και με ένα περιορισμένο μέγεθος γνωμοδότησης γιατί είναι δεδομένο αυτό. Πριν από λίγε εβδομάδε ενημέρωσα του κοιοδησηγητέ για τα εξή θέματα. Πρώτον, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει πρόθεση αναθεώρηση του Μητρώου Διαφάνεια στα πλαίσια ε, τη ευρύτερη ε, και συμμετοχική ε, δυνατή διαβούλευση. Επίσης, να συνεχίσει τι συζητήσει για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ομάδα χωρών κατά τη διαφθοράς. Επίσης, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει γνωμοδότηση για τους καταγγέλλοντες whistleblowers από το 2016 και μετά. Ανεξάρτητο γραφείο εισαγγελέα και δυνατό για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και μάλιστα το συντομότερο. Επίσης, και την απάτη κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους για την πρόσβαση στα έγγραφα και να βελτιώσουμε ε, την διαφάνεια των νομοθετικών διαδικασιών συμπεραμαλωμένων δε και των τριμερών διαλόγων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνούν και οι σκιώδεις που τους ρώτησα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Ε, να δημιουργηθούν οι αρμόδιες αρχές για τη διαφάνεια, τα κράτη-μέλη ανθίστανται ακόμα, ε, να γίνονται έλεγχοι ε, για τις πληροφορίες που ε, γράφονται στο Μητρό. Ξέρω ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και των ισχρών αγελάδων δεν θεωρούν προτεραιότητα, αλλά στο πούμε. Και επίσης να καταλαβαίνουν οι πολίτες τι γίνεται για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, ότι κάνουμε αυτές τις προσπάθειες και τις πολιτικές και να δείξουμε στους πολίτες ότι καμιά φορά οι βουλευτές τους μπορεί και αυτοί να αμφιβάλλουν και να αμφιταλαντεύονται. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά αυτή είναι μόνο ένα στοιχείο της λύσης του προβλήματος. Υπάρχει μια διαδικασία πιο μακροχρόνια που σημαίνει ότι χρειάζεται εις βάθος αλλαγή και των νοοτροπιών και των ε, αντιλήψεων για να δώσουμε το καλό παράδειγμα κάθε εκλεγμένος έχει και μια ηθική ευθύνη, αλλά υπάρχουν και όρια, τα όρια της λογικής. Και ένα τελευταίο θέμα, δεν θα πρέπει να συμβάλλουμε στο να ε, καλλιεργούμε ένα κλίμα γενικευμένης καχυποψίας για τους πολιτικούς, που αυτό είναι νερό στο μήλον των λαϊκιστών και μόνο ελπίζω να καταλήξουμε ε, στην κατάλληλη ισορροπία για το θεσμικό μας όργανο και για τους πολίτες, τους οποίους εμείς πάντα πρέπει να λογοδοτούμε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Σιλβί. Άλλος συνάδελφος που θέλει το λόγο. Η Ρομπέρτα Μετσόλα. Claude, um, I'm... Ευχαριστώ, Κλοντ. Και μου ζήτησε ο κ. Τεχόφσκι να ο εξ ονόματός του για το θέμα αυτό. Μπορώ να πάρω το λόγο τώρα. Πολύ ωραία. Εξ ονόματος λοιπόν του Τόμας που ήταν σκιωδής του ΕΛΚ θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Κιγιόμ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Το σχέδιο περιλαμβάνει όλα όσα συμφωνήθηκαν σε επίπεδο σκιωδών. Ωστόσο, ο κ. Τεχόφσκης θεωρεί ότι η έκθεση είναι υπερβολικά γενικόλογη και είναι προς το συμφέρον της Επιτροπής μας να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και ισχυρή γνωμοδότηση για το θέμα αυτό, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο το Κοινοβούλιο, αλλά όλη τη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια στα θεσμικά όργανα και πιστεύουμε ότι το υποχρεωτικό μητρό για τα λόμπι, για τη διαφάνεια, το οποίο εισήγαγε και ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο Τίμερμαντς ε, στην ε, στο Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ, πολύ σύνθετο. Σε ό,τι αφορά τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers, ε, συμφωνεί ο κ. Δουχόφσκι ότι χρειαζόμαστε ελάχιστους κανόνες για την προστασία τους, αλλά θα πρέπει να τύχουν σωστή συζήτηση οι κανόνες αυτές. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του τρομερού διαλόγου, θα ακολουθήσουμε τις συστάσεις του κυρίου Σούλτς που επεσήμανε ότι πρόκειται για μια εμπιστευτική διαδικασία που δεν μπορεί να μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η κατάσταση των διαβουλεύσεων θα πρέπει να ε, ανακοινώνεται τακτικά στην Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφάνειας και το θέμα της ε, εκλογής και του διορισμού των διευθυντών και των υποδιευθυντών στο πλαίσιο αυτό. Θα τονίσουμε και αυτό. Τέλος η ομάδα του ΕΛΚ πάντα αναζητά τη σωστή ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και προστασίας δεδομένων και αυτό θα το κάνουμε και στην τρέχουσα γνωματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει προεδρό Πρόεδρος, Ρομπέρτα. Αν, άλλο ένα μέλος έχουμε, την Άννα Γκόμες που θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ καλωσορίζω ιδιαίτερα τη γνωμοδότηση αυτή και πιστεύω ότι πραγματεύεται και κάποια κρίσιμα ζητήματα. Εκεί θα πρέπει να επιδείξουμε όσο πιο μεγάλη ακρίβεια γίνεται. Και το θέμα της διαφάνειας ασφαλούς. Στο μήτρο των λόμπι. Η προστασία των ε, καταγγελόντων. Είναι ένα βασικό ζήτημα και αυτό. Για τη διαφάνεια των ε, τριμερών διαλόγων. Όντως, θα συμφωνήσω ότι δεν είναι ενδεχομένω ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων. Γιατί αν υπάρξει πλήρη διαφάνεια, πολύ απλά θα φύγουν οι διαβουλεύσεις από την πλατφόρμα αυτή. Και ανησυχώ ιδιαίτερα και για διάφορες υποθέσεις ε, διαφθοράς κυρίως. Τις έχω θέσει και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την Όλαφ. Τις έχω καταθέσει και στην Διαμεσολαβήτρια και θα πρέπει να σας πω ότι το μοναδικό θεσμικό όργανο που απαντάει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας. Γιατί πραγματικά από πλευράς Επιτροπής τα πράγματα είναι τραγικά. Και αυτό είναι άλλος ένα λόγος που με οθεί στο να λέω ότι θα πρέπει να επιδείξουμε όσο πιο πολύ ακρίβεια γίνεται στην έκθεση αυτή με συγκεκριμένες υποθέσεις. Και ανησυχώ γιατί η επόμενη έκθεση για την διαφάνεια πολύ φοβάμαι θα ακολουθήσει το μονοπάτι της ε, παλιάς. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι πολλές από τις υποθέσεις που έχουν επισήμανθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάληξαν σε υποσημειώσει. και δεν συμπεριλήφθησαν και τελικά δεν έγινε και τίποτα. Είναι θλιβερό και απαράδεκτο. Απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει και αυτό το λέω ιδιαίτερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν πολλά κέρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είχα μεγαλύτερε προσδοκίε. Είχα τι πιο υψηλέ προσδοκίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και απογοητευτήκαμε έκτρα και με την προηγούμενη επιτροπή. Αλλά συνεχίζεται και αυτή η παράδοση στη σημερινή επιτροπή και στην αδράνειά της σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις διαφθοράς τις οποίες έχω επισημάνει και εγώ και άλλοι στην Επιτροπή. όχι μόνο της ε, αμελή, αλλά της, ε, σχεδόν της καλύπτει, της συγκαλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποδέχεται διάφορες δικαιολογίες από τα κράτη-μέλη. Ο Πρόεδρος δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο να ζητήσω από τη Σιλβή να μας πει κατά πόσον θέλει να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή προτιμάται όχι. 22 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες να απαντήσω να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα απαντήσω και εγώ στους συναδέλφους. Μάλιστα. Και η συγγήτρια λοιπόν θα ήθελε να ακούσει δύο λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Some uh, Αν θέλετε να σχολιάσετε. Δεν ε, μπορείτε ίσως να επισέλθετε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας. Αλλά αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω εκ νέου ότι η Επιτροπή Juncker τονίζει όλος ιδιαίτερος τα θέματα αυτά τα τονίζει λοιπόν, ακεραιότητα, διαφάνεια και είναι ύψιστη προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Juncker αυτά. Διαφάνεια, η ακαιρεότης έχει διάφορες οπτικές γωνίες και πρέπει να ακολουθήσουν ε, διαφορετικές διαδικασίες, να ακολουθηθούν. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε σε σημαντικότατα θέματα που σχετίζονται με αυτά. Προφανώς όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα θα θέλαμε να δούμε πώς αυτά εντάσσονται στη γενική έκθεση, στο τελικό κείμενο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δέσμευση να απαντήσει επισήμως από αυτόν ε, εντός της διαδικασίας της συνεχείας που θα δοθεί θα θέλαμε να στηρίξουμε τη θέση σας στο μέτρο του δυνατού. Σαφής πρωτοβουλία, σαφής προτεραιότητα πρωτοβουλίας της Προεδρίας είναι να γίνει το Μητρό υποχρεωτικό. Και θα πρέπει να πετύχουμε τριμερή διοργανική συμφωνία από αυτό. Όπως γνωρίζετε άλλες στοιχεία διαφανείας καλύπτονται σε άλλους τομείς. Όπως η καλύτερη, η καλύτερη νομοθεσία του θετικού πακέτο και η δέσμευση που αναλάβουμε περί αυξήσεως διαφανείας, ομάδες εμπειρογνωμόνων κλπ. Αυτή είναι η γενική μας άποψη. Για τις εικασίες που ακούστηκαν από την κυρία Βουλευτή για τη λειτουργία της ΟΛΑΦ. Ερήτημη κυρία, δεν γνωρίζω την ε, ακριβή αυτή περίπτωση. Όποτε ενδεχομένως υπάρξει λόγος επανεξετάσεως διενεργηθισών αξιολογήσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά χαράς να το κάνουμε. Πρέπει να κατανοήσετε ότι έτσι αφηρημένα δεν μπορώ να σχολιάσω διότι οι κασίες αυτές, οι κατηγορίες αυτές ήταν, οι καταγγελίες μάλλον, οι κατηγορίες ήταν πολύ αόριστες. Σιλβί. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σημειώνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα το γεγονός ότι ε, αρκετές προοπτικές ε, παραμένουν ενισχύ. Ωραία όλα αυτά, ε, να τους δώσουμε κάπως σάρκα και ωστά. Υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρό, δεν το είχα καταλάβει ότι ήταν η πρόθεσή σας τόσο το καλύτερο. Για τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, να απαντήσω ότι βεβαίως όλες οι τροπολογίες ε, είναι ευπρόσδεκτες για να διαρθρωθεί αυτό το κείμενο που είναι πάρα πολύ περιορισμένο γιατί έχουμε περιορισμό στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνταχθεί η γνωμοδότηση να παραμείνουμε όμως στα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, της Επιτροπής Ελευθεριών. Η έκθεση είναι του συναδέλφου Γκίγκολτ. Είναι πολύ συγκεκριμένη και εκεί ασχολείται με όλα τα θέματα. Εμείς να δούμε τα δικά μας ζητήματα. Για το θέμα των κατακελώντων που είπε η κυρία Γκόμες, η παράγραφος 44 σε αυτό αναφέρεται. Και σας ευχαριστώ την προσοχή για τους whistleblowers και είναι και προς την κατεύθυνση που εσείς θέλετε. Ευπρόσδεκτες οι τροπολογίες καλώς να ορίσουν, να περιοριστούμε στα θέματα της ΛΥΠΕ και να φροντίσουμε να έχουμε όσο πιο ακριβή και λεπτομερή ε, γνωμοδότηση γίνεται. Ευχαριστώ. Ωραία συμβουλή αυτή να επικεντρωθούμε στα θέματα της Επιτροπής μας και να περιοριστούμε σε αυτά. Ε, γιατί πιέζει και ο χρόνος για την κατάθεση των τροπολογιών. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι και εσένα Σιλβί. Yeah, no, that. Okay, colleagues, Σημείο 6 είναι το επόμενο βέβαια. Διαρθρωμένος διάλογος με τη Βέρα Γιώροβα. Ε, κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, ένα διάλειμμα, να περιμένουμε την κυρία Επίτροπο. Πηγαίνετε να πάρετε κανένα τσάι.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 colleagues, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να έρθει η Επίτροπος. Είναι και πέμπτη, τώρα τα ξέρουμε ε. αυτά, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Παρακαλώ να επιστρέψετε αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σε πέντε λεπτά πάνω κάτω.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 Um, colleagues, um, I uh, Αδελφοί, πέρασε το πετάλεπτο. Έχει έρθει ο Επίτροπος. Θέλω να τσεκάρω. Ε, έκανα λάθος εγώ γιατί έκανα διάλειμμα και είπα στον κόσμο να πάει για καφέ. Εγώ καφέ βέβαια πήρα, αλλά πού είναι. εδώ σε αυτά τα κτίρια έτσι όπως έχουμε καταντήσει ότι για καφέ δεν μπορείς να πας μέσα σε πέντε λεπτά. Τα πάντα χρειάζονται από τέταρτο και πάνω. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε στους συναδέλφους σας ότι έχει έρθει επίτροπος παρακαλώ και στους ε, βουλευτές σας και τα λοιπά. Είναι έτοιμη η επίτροπος εδώ και έχει έρθει να συζητήσει μαζί μας. Α, θέλει και καφέ. Καλά. Ε, χάσατε όμως, αργήσατε. Άλλο θεσμικό όργανο ε, εκείνοι. Όταν θέλουν καφέ τους φέρνουν. Θα ξεκινήσω λοιπόν συνάδελφοι. Στείλτε κανένα μήνυμα στους συναδέλφους να έρθουν γιατί πέρα από τα στιάκια τώρα είναι σημαντικό το θέμα και θέλουμε να το κουβεντιάσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που λείπουν και θέλουν να ξανάρθουν. Μήπω αυτή την ε, προϋπόθεση, αυτή τη συνθήκη κλπ. Να ξεκινήσουμε, τι λέτε. Καλώ. Είναι πέμπτη και κάποιοι έχουν να ταξιδέψουν. Ας ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την υπομονή σας. Συνάδελφοι, σημείο 6, διαθρωμένος διάλογος με την Επίτροπο κυρία Γιουρόβα, κάτι που υποσχεθήκαμε σε όλους. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα που ε, ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό της. Είχαμε πει όμως και το συζήτησαν και οι ότι θα μιλήσουμε για περαιτέρω πληροφορίες για τον ασφαλή λιμένα, το Safe Harbor και τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ. με αυτή τη συντομότερη από ό,τι συνήθως εισαγωγή. Θα ζητήσω από τη Βέρα Γιουρόβα να πάρει το λόγο. Βέρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ ξανά. Για το διαστρωμένο διάλογο μαζί σας, για τα διάφορα ζητήματα και τα θεματολόγια κοινού ενδιαφέροντος και είναι καλή σύμπτωση το ότι σήμερα μπορούμε μαζί να γιορτάσουμε τη Διεθνή ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η επέτειος του, της συμβάσεως του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1950. Έχουμε λοιπόν αυτή την ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου που είναι πολύ συμβολική και για τη συνεργασία μας στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε έναν κατάλογο δράσεων που θέλει να προωθήσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Αυτό το παρουσίασα στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα. Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστώ θέρμα την Αντιπρόεδρο Λούνατσεκ. Είναι εδώ. Ναι. Όχι, όχι δεν είναι. Εδώ ήταν. Ίσως έρθει. Διαβιβάστε λοιπόν τις θερμές μου ευχαριστίες και χαιρετίσματα. Διότι σαν πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ομάδας για τους ΛΟΑΔ μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και ήταν άριστη η συνεργασία μας εν την επεξεργασία του καταλόγου. Οι δράσεις καλύπτουν πλήρως βασικούς τομείς πολιτικής για τους ε, ΛΟΑΔ. Μη διάκριση συμπεριλαμβάνεται. Παιδεία, απασχόληση, υγεία, ελεύθερη διακίνηση, άσυλο, καταπολέμηση κατά μυσαλλοδόξων λόγων και εγκλημάτων μυσαλλοδοξίας, εξωτερικές σχέσεις κλπ όπως βλέπετε στον κατάλογο, ο οποίος έχει διανεμηθεί, να τος αυτός εδώ είναι. Αρκετά πολύχρωμος. Μπορείτε να δείτε στον κατάλογο ότι επιμένουμε επί της σημασίας της εγκρίσεως από το Συμβούλιο ε, κρεμουσών προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου που έχουν σημαντική και άμεση συνέπεια για τους ΛΟΑΔ όπως ισότιμη αντιμετώπιση που περιέχεται στην σχετική οδηγία. Είναι μια νομοθετικού περιεχομένου πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ολοκληρωθεί του χρόνου. Έχω άριστη συνεργασία με την επερχόμενη Ολλανδική Προεδρία που θα δώσει και αυτή η Προεδρία ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θέμα. Ταυτόχρονα επιβολή των μέτρων, εφαρμογή της υφισταμένης νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Αν γίνουν όλα αυτά θα ωφεληθούν οι ΛΟΑΔ. Θα προστατευτούν καλύτερα. Παρακολουθούμε σε συνεργασία με τα κάτι μέλη την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αρχή της μη διάκρισης θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ισχύει και εφαρμόζεται συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτυχών που αφορούν το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα όσον αφορά το φύλλο. Λοιπόν, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια θα παράσχουμε οικονομική ε, στήριξη, ηλεκτρονική εκμάθηση, e-learning και κατάρτιση σε εκείνους που δίνουν ίσα δικαιώματα στους ΛΟΑΔ και στα κράτη-μέλη, στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες των πολιτών. Πρέπει να πλησιάσουμε τους πολίτες και να γίνουν πιο αποδεκτοί από τους πολίτες οι ΛΟΑΔ. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μου. Θα ξεκινήσω ε, μια εκστρατεία το 2016 όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ευαισθητοποίηση Εκεί θα πηχούνται οι ανησυχίες των πολιτών μας που είναι ΛΟΑΔ. Θα ζητούμε ανοχή, σεβασμό και θα τονίσουμε και το πόσο καλό είναι να υπάρχει ποικιλομορφία στην κοινωνία. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας. Να γίνετε πολλαπλασιαστές στις χώρες σας αυτών των μηνυμάτων. Όσον αφορά την μεταρρύθμιση για την προστασία των δεδομένων, έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε πολιτική συμφωνία εφέτος κατευθυνόμεθα προς ε, κρισίμους τριμερείς διαλόγους αυτή την εβδομάδα και θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στο έργο των εισηγητών, των κυρίων Άλμπρεχτ και της κυρίας Λορεστίν και των σκιωδών εισηγητών. Διότι ηγήθηκαν στις προσπάθειες. Χάρη στις δικές σας προσπάθειες και στις προσπάθειες των διαδοχικών προεδριών του Συμβουλίου και της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας πιο συγκεκριμένα έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος του έτους. Γράφουμε ιστορία ολοκληρώνοντας τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων. Ο κανονισμός μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε την ενιαία ψηφική αγορά. Έχουμε κοινού κανόνε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι κρισίμου σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη στην παγκόσμια οικονομία. Οι νέοι κανόνε επίση θα προωθήσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα προωθήσουν. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η οικονομική ανάπτυξη πάνε χέρι με χέρι. Είμαι, έχω την πεποίθηση ότι οι επιτευχθεί σε συμφωνίε των τριμερών διαλόγων θα εξασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία των ατόμων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες που θα προσφέρει η ψηφιακή οικονομία και θα αντιδικοποιηθεί η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί και θα είναι φιλική όσον αφορά την προστασία την, ε, της ιδιωτικής ζωής. Και η οδηγία σχετικά με την αστυνόμευση είναι σημαντική για το όλο θέμα της ε, ασφαλείας. Κοινοί κανόνε για την ε, προστασία των δεδομένων θα επιτρέψουν δικαστικές αστυνομικέ αρχέ να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα μεταξύ του και μια συμφωνία επί του χαρτοφυλακίου είναι ακόμα πιο πιεστική τώρα μετά από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις εις Παρισίους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένε Πολιτείε για τον ανωμένο πλαίσιο για τη διατλαντική ανταλλαγή στοιχείων. Οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τώρα που μιλάμε, ο στόχος μου παραμένει να δημιουργήσουμε μια δομή που θα έχει οδηγήσει σε πιο ε, ισχυρό σύστημα εποπτείας και ελέγχων. Έχουμε καθορίσει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των συνομιλιών και παραμένω αισιόδοξη. Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή βεβαίω ότι θα πληρούνται οι κατάλληλε προδιαγραφές. Επανειλημμένα έχω τονίσει όταν μιλούσα με τους συνομιλητές μου στη ΣΥΠΑ και στην επίσκεψή μου την πρόσφατη στην Washington DC μέσα Νοεμβρίου ότι πρέπει να συνεργαστούμε σκληρότερα για να τα καταφέρουμε. Η ΕΠΑ θα πρέπει να δείξει κατανόηση ευελιξία και δημιουργικότητα ώστε να βρεθούν αξιόπιστες ε, λύσεις. Το χρωστούμε σε επιχειρήσεις μας και τους πολίτες. Οι νέες διευθετήσεις θα πρέπει να είναι σταθερές και βιώσιμες. Ένα θέμα το οποίο συζητούμε είναι το πώς οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά εποπτεύοντας τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις νεδιαθετήσεις. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε το σημαντικό ρόλο των διαφόρων αυτών σημαντικών ε, των εποπτικών αρχών στην απόφαση ΣΡΕΜΠΣ και θα πρέπει να εποπτεύουμε το πλαίσιο μέσω των αρμοδίων αρχών των χωρών μας ή σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ με την Ομοσπονδιακή Αρχή Εμπορίου που θα πρέπει να εφαρμόσει τις κατάλληλες υποχρεώσει, να υλοποιήσει κατάλληλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, θέλουμε αποτελεσματική εποπτεία και να υπάρχει δυνατότητα ε, οι, οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη όταν αυτόν παρίσταται αναγκαίο στον αφορά την χρήση των δεδομένων του. Θέλουμε περαιτέρω διαβεβαίωση από τη ΣΥΠΑ ότι η πρόσβαση από τι δημόσιε αρχέ για λόγου εθνική ασφαλεία από τις αρχές ασφαλείας και για σκοπούς δημόσιας ασφαλείας θα είναι περιορισμένη πρόσβαση μόνο όσο είναι αναγκαία. Και αναλογική πρέπει να είναι, θα πρέπει να τίθενται ρήτρες διαφύλαξης και περιορισμοί, θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για δικαστικό έλεγχο, δυνατότητα αποζημίωσης, ε, συνθήκες χρήσεως των στοιχείων κλπ ε, και κυρίως για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αυξήσουμε την, τις αναφορές όσον διαφάνεια, όσον αφορά τα αιτήματα για πρόσβαση από τις δημόσιες αρχές, ούτω ώστε να αποδεικνύεται ότι οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας εφαρμόζονται επίσης στην πράξη. Η αδίποτε νέα αρρύθμιση θα υπόκειται σε αιτήσει αναθεωρήσεις και ελέγχους. Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή για να σας διαβεβαιώσω ότι μετά τις επιθέσεις εις Παρισίου στις 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση ε, του ξεπλήματος χρήματος και νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και την καταπολέμηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Με την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, έχουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να εντοπίζουμε καλύτερα και να ανοιχνεύουμε, να ανοιχνεύουμε την προέλευση δισεκατομμυρίων ε, ευρώ που προέρχονται από οικονομικές απάτες και από παράνομες δραστηριότητες που υποστηρίζουν παράνομες ομάδες στις δραστηριότητες. Θέλουμε ταχεία και αποτελεσματική ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και τα κράτη-μέλη υποσχέθηκαν ότι θα επιταχύνουν την εφαρμογή αυτή. Εγώ έχω αναλάβει να εντοπίσω και να προτείνω περαιτέρω μέτρα που είναι κατάλληλα για να καταπολεμήσουν την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε την απάντησή μας και τη συνεργασία μας με άλλους διεθνείς εταίρους μας. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν του θεματολογίου για την ασφάλεια ε, θα επιταχύνουμε επίσης τις εργασίες επί του ΕΚΡΙΣ που είναι το μητρό όσον αφορά το, το ποινικό μητρό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα παρουσιάσουμε μία επέκταση του συστήματος ανταλλαγής ποινικών μετρών σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτό θα είναι σημαντικό εργαλείο στην αποτελεσματική διασυνοριακή επιβολή του νόμου και στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως είναι και η τρομοκρατία. Η επόμενη, η Ολλανδική Προεδρία, ε, προοδεύει τάχιστα στο σημαντικό αυτό χαρτοφυλάκιο. Θα επανέλθουμε επ' αυτού στο επόμενο Συμβούλιο μετά το νέο έτος. Επίσης προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου ε, στο, όσον αφορά το θέμα της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Η PPO θα το αποκαλώ από τώρα σύντομα. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει εν γέννη υποστήριξη όσον αφορά ένα θεωρημένο κείμενο που θα διέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εγγελίας δομή φερρυπίν, αρμοδιότητες, μέτρα ερεύνων και διάφορα δικαιώματα για τις διαδικασίες που μπορεί να ακολουθεί. Τίποτα όμως δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι συμφωνηθούν όλα. Είμαι αποφασισμένη να έχουμε το 2016 μία ανεξάρτητη ε, εισαγγελία και οι επόμενες προεδρίες, η Ολλανδική και η Σλοβακική, είμαι σίγουρη ότι θα ασχοληθούν με τα κρεμή ζητήματα και θα ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαπραγματεύσεις. Να τονίσω εκ νέου. Το Κοινοβούλιο διαδραματεί σημαντικό ρόλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άκουσα τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, καθώς και αυτές που εκφράστηκαν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήσασταν σαφείς στις δύο διάμεσε εκθέσει. και συμφωνώ με πολλές από τις ανησυχίες σας και θα καλωσόριζα την ισχυρή φωνή του Κοινοβουλίου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα όσον αφορά την οδηγία κατά καταπολεμήσεως της απάτης, θα πρέπει να βρούμε κάποιο συμβιβασμό όσον αφορά τη συμπερίληψη του ΦΠΑ. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην Τράπεζα των Υπραγματεύσεων τώρα και να τονίσουμε το πόσο σημαντικές είναι οι ληφθήσεις αποφάσεις του δικαστηρίου. Εάν εξαιρούσαμε το ΦΠΑ θα ήταν ένα βήμα επαναχώρησης και όχι πρόοδου και θα ήταν αντίθετο με το στόχο της οδηγίας, δηλαδή να ενισχυθεί το επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ενώσεως. Τώρα, σχετικά την συνεργασία στο δικαστικό τομέα, να υπογραμμίσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν με καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα που προσφέρει το Eurojust και τα σχετικά εργαλεία. Παραδείγματο χάρη διευκόλυνση των ερευνών και των διώξεων, κοινέ ερευνητικές ομάδες, συνεδριάσεις συντονισμού και συνεργασία με τρίτες χώρες, κυρίως με χώρες μήνα και των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και τέλος, ας δούμε ποια είναι τα διάφορα ε, δικαιώματα δικονομικά δικαιώματα. Κυρίω για τα παιδιά ε, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλο του έτου οι διαπραγματεύσει. Για να φτάσουμε σε τελικό συμβιβασμό θα πρέπει να βρούμε ένα ισορροπημένο κείμενο όσον αφορά τη βοήθεια που μπορεί να παράσχει νομικό στα παιδιά. Η παροχή νομικής αρρωγής στα παιδιά είναι βασικό στοιχείο της οδηγίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους ή όπου η στέρηση της ελευθερίας θα μπορούσε να επιβληθεί ω κύρωση χρειάζεται να καθοριστούν ε, πολύ στενοί περιορισμοί και να είναι πολύ σαφώς καθορισμένα τα όρια. Είναι σημαντικότατο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει συμφωνία στο εγγύς μέλλον όσον αφορά την οδηγία περινομικής αρρωγής, ούτως ώστε το δικαίωμα, στην πρόσβα... πρόσβαση στον νομικό να λειτουργεί. Η οδηγία της πρόσβασης στην νομική αρρωγή θα πρέπει να σωματωθεί στα εθνικέ σε εθνικές νομοθεσίες μέχρι 27 Νοεμβρίου του 2016 χωρίς να συμπληρώνεται με ένα στέρεο δικαίωμα για νομική αρρωγή, υπάρχει κίνδυνο στα δικαιώματα που προβλέπει η οδηγία να παραμείνουν κενό γράμμα. Για να απεμπλακούν οι διαπραγματεύσεις απαιτείται ευελιξία από την πλευρά του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά βασικές διατάξει της οδηγίας είναι κάτι που προτάθηκε από τον εισηγητή τον κ. Ντεγιόν και πρέπει να ξεκινήσουν αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει τι προτάσει του Ευρωκοινοβουλίου για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία, όσον αφορά την νομική αρρωγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει τον εισηγητή ο οποίο έχει δρομολογήσει μια αξιολόγηση συνεπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζει ότι αυτή η έκθεση θα είναι διαθέσιμη το ταχύτερον δυνατόν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πολλά θέματα και καλό θα είναι να έχουμε το χρόνο να επεκταθούμε σε αυτά. Θα πάμε αμέσω στους ομιλητές με πρώτη την κυρία Χόλμαϊερ που πήγε. Έρχεται. Έλα. Αυτά είναι. Ψηφίσαμε και φύγαμε μπαινοβγαίνει ο κόσμος και μετά αυτά παθαίνουμε. So, um, επιστρέφω, θα τους δίνω το λόγο. Η Μπίρκη Τσίπελ είναι παρούσα, έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπό μας που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας. Καμιά φορά ανησυχούμε ε, όλοι όταν βλέπουμε μικρή παρουσία βουλευτών. Αλλά όπως είπε ο Κλοντ, σε κάτι διαφορετικό οφείλεται αυτό. Χαίρομαι που λέει η Βέρα Γιούροβα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν καλύτερα όχι μόνο τη Europol αλλά και τη Eurojust. Να συνεργάζονται καλύτερα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται και έχει σημασία τέτοιες μέρες αυτό, όταν πρόκειται για τη διαφθορά και την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω εδώ επίσης τη σημασία του να έχουμε ένα ισχυρό Ευρωπαίο εισαγγελέα, Ευρωπαϊκή εισαγγελία, Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη, αλλά να καταλάβουν ότι πολλή δουλειά έχουν ακόμα να κάνουν και στα κράτη γιατί υπάρχουν προβλήματα καταχρήσεις ε, χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να φτιάξουμε άντε μια εισαγγελία ευρωπαϊκή, όχι. Να έχει ε, ισχυρές αξιωσίες και αρμοδιότητες δράσης σε αυτό το τομέα ε, της διασπάσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι είναι καλή η συνεργασία στο ποινικό δίκαιο σε θέματα που εκκρεμούν ακόμα το συμφέρον των παιδιών και η νομική ε, αρρωγή. Επίσης χαίρομαι που υποστηρίζετε την ιδέα να υπάρξει μια μελέτη αντικτύπου ε, και επιπτώσεων για να δούμε που υπάρχουν κενά παραθυράκια και ελλείψεις και να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα με τα κράτη-μέλη πάντα στη συνεργασία. Να σας ρωτήσω για τον ασφαλή λιμένα, το λεγόμενο Safe Harbor. Γιατί έχουμε το εξή πρόβλημα. level, Ε, η διαπραγμάτευση γίνεται σε εθνικό επίπεδο ε, και έχουμε διαφορές και στα κράτη-μέλη αλλά και στις ΗΠΑ από πολιτεία σε πολιτεία. Δεν είναι όλα αυτά ε, ίδια. Πώς λοιπόν θα καταλάβουμε ε, σε ποιο επίπεδο γίνεται οι συνομιλίες και ποιο επίπεδο κυριαρχεί. Σε εμά είναι σε κρατό ε, μελών, στις ΗΠΑ είναι αναπολιτεία ή στο σύνολο της χώρας. Επίσης, πώς θα υπάρξει κάποιο στοιχειώδης έλεγχος σε μπάση περιπτώσει, ότι όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι φορείς συμμορφώνονται με κάποιους κανόνες που έχουν συμφωνήσει προηγουμένως. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω Μπορείτε προς το παρόν να μας πείτε τι γίνεται από πλευράς χρονοδιαγράμματος, πότε διαβλέπετε έτσι κάποια συμφωνία από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπίργκιτ. Ο κύριος Κύρκοπ, επόμενος συντονιστής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρία γρήγορα σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Απουσία οδηγίας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Τι μέτρα πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει και να ε, εξασφαλίσουν ε, την προστασία των δικαιωμάτων χωρίς ε, νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Ανησυχώ σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την ταχύτητα των μέτρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προγραμματίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στη φάση της εφαρμογής. Και μία ερώτηση να κάνω από πλευρά τη κυρία Μάκοβε, εξ ονόματο τη συναδέλφου. Θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με τις ε, διαπραγματεύσεις για το EPPO μετά το τελευταίο συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα θέλει να ρωτήσει τι γίνεται με τα βασικά ζητήματα για τον Εθνικό Σύνδεσμο και την αναγνώριση των κρατών μελών και που θα έχει δικαιοδοσία η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εισαγγελία. σε ό,τι αφορά την εισαγγελία, λοιπόν. Μάλιστα. Η κυρία Σαρτζεντίνη, λέει ο πρόεδρο, είπαμε στην Ιστρία. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν θα κάνω όλε τι ερωτήσει ε, που φαντάζομαι ότι θα έχουν απαντηθεί. Ένα συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να θίξω. Αυτό εδώ. Αυτέ οι δράσει, ο κατάλογο δράσεων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθηθεί η ισότητα των ΛΟΑΤ και εξ ονόματος της συνάδελφου Λούνατσεκ. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς ερμηνεύεται αυτός ο τίτλος «Κατάλογος δράσεων», «List of Actions». Αυτό δεν είναι δεσμευτικό για όλη την Επιτροπή, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Ίσως μόνο για την Επίτροπο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται και κατά πόσον είναι δεσμευτικό και πώς. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα γίνει η υποβολή εκθέσεων βάσει των ε, δράσεων αυτών, από ποιον και προς ποιον. Για μας τους πράσινους είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθεί ο δικός χάρτης για την ισότητα των ΛΟΑΔ. Ευχαριστούμε, Τζουντίθ. Η κυρία Κορατσαμπίλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελε να σας ευχαριστήσω ε, Επιτροπέ, για την εξαιρετική συνεργασία, την εξαιρετική, διαθεσιμότητα, τον εξαιρετικό διάλογο του τελευταίο χρονού. Να σας συγχαρώ επίσης για την έκθεση, για τον κατάλογο δράσεων για την ισότητα των ΛΟΑΤ. Μιλήσατε για την οδηγία για την ίση αντιμετώπιση. Είμαι σκιώδης από πλευράς ε, του ΕΛΚ. Και όπως ξέρετε στο Συμβούλιο έχει μπλοκάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό η οδηγία κατά των διακρίσεων. Και ελπίζω να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να κάμψετε την πολιτική αντίσταση και για να είμαι πιο α, συγκεκριμένη. Τι κάνετε για να επιβάλλετε πίεση στο Συμβούλιο. Είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονό ότι καθυστερεί τόσο πολύ η νομοθεσία για την κατάργηση των διακριτικών μεταχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ασφαλή λιμένα, είπατε και εγώ απογοητεύτηκα ιδιαίτερα από τις δηλώσεις του κυρίου Τίμερμανς και τις δικές σας, και τις δικές σας δηλώσεις μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Χιλιάδες ε, τέτοια δεδομένα, χιλιάδες ε, επιχειρήσεις δεν έχουν την νομική βεβαιότητα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Αυτό επηρεάζει την ελεύθερη ροή των δεδομένων που αποτελεί μία από τις βασικές ε, ελευθερίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι υπέρ της προστασίας ε, των δεδομένων, αλλά χρειάζεται τάχιστα νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα και οι κατευθυντήριες ε, γραμμές τις οποίες δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο πολύ απλά δεν αρκούν. Ελπίζω λοιπόν να προωθηθεί η εργασία αυτή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ροή των δεδομένων αυτών. Ένα τρίτο σημείο. Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Όπως ξέρετε, καταρτίζουμε μια έκθεση, εφαρμοστική έκθεση για τον κανονισμό του 2001 και είμαι σκιώδης από το ΕΛΚ. Αλλά και πάλι, ο νέος κανονισμός που αναβαθμίζει και δίνει πιο πολλές ευκαιρίες διαφάνειας στους πολίτες, έχει μπλοκάρει και δεν κινείται εδώ και πολύ καιρό. Τι προτίθεστε λοιπόν να κάνετε για να προχωρήσει το θέμα αυτό, κυρίως στο Συμβούλιο αλλά και στην Επιτροπή. Τελευταίο θέμα, για τα παιδιά. Χάρηκα που αναφέρατε το, αναφέρθηκε το θέμα της αρρωγής ε, των δικηγόρων προς τα παιδιά στην έκθεση Κινίτσι. Και το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει μια νέα ατζέντα για τα παιδιά. Μια και εκμηνέει το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, είχε ανακοινώσει ότι δεν ε, σκόπευε να προτείνει μια νέα ατζέντα. Τι είδου μέτρα λοιπόν, τι είδου δουλειά θα προγραμματίσετε για τα επόμενα πέντε χρόνια για να υπάρχει μια στρατηγική εναρμόνιση των δράσεων για τα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γλώμπας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Γιώροβα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτό το διαρθρωμένο διάλογο και που μας δίνετε την ευκαιρία να έχουμε διάλογο ουσιαστικό με θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Κάνατε λόγο για την κατάσταση των πραγμάτων, ε, για την οδηγία προστασίας των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνεργασία σε ποινικό επίπεδο. Πολύ σύντομα αναφερθήκατε έτσι επιγραμματικά στις τελευταίες συζητήσεις και μάλιστα την πιο πρόσφατη στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων πριν από λίγες μέρες. Θα ήθελα όμως να μάθω ε, τι χρονοδιάγραμμα προβλέπετε εσείς για αυτά τα θέματα. Πότε αναμένετε να έρθουν. Πότε θα απεμπλακεί όλο αυτό το θέμα που είναι φρακαρισμένο για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Γιατί γίνεται ένας πόλεμος για το ΦΠΑ από ό,τι έχω καταλάβει. Είχαμε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κάποια ισορροπία πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή και κάπου να συναντηθεί το Συμβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιες γέφυρες πρέπει τώρα να χτιστούν έτσι ώστε επιτέλους να καταλάβουμε ότι το ΦΠΑ είναι ένας πόρος για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ίδιος πόρος που δεν προϋποθέτει ε, την αρμοδιότητα που επικαλούνται τα κράτη-μέλη για θέματα φορολογικά. Επίσης, αυξάνεται η ανησυχία για την έξαρση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και μας προβληματίζει, μας έχει ανησυχήσει πάρα πολύ ε, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία είναι θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ο αντισημιτισμός ιδιαίτερα στην Ουγγαρία. Θέλω να μάθω Έχετε ακούσει για μια περίπτωση γιατί εγώ είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας κατά τον συμβιτισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενημερωθήκαμε ότι σε ένα ουγγρικό χωριό που λέγεται Ζέκες Φερχερβάρα, κάπως έτσι και ζητώ συγγνώμη για τα ουγγρικά μου. Σε αυτό το χωριό λοιπόν πρόκειται να στηθεί ένα μνημείο στη μνήμη του Μπάλιτ Χόναν που ήταν πρώην υπουργό της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης στη δεκαετία του 30 και του 40 που συμμετείχε ενεργά στην έγκριση αντι-Ισραηλιτικών νόμων και που ευθύνεται για τους εκτοπισμούς εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων. Ουγγρό Εβραίων στο ολοκαύτωμα. Το έχετε ακούσει αυτό, το έχετε υπόψη σας και αν σας ανησυχεί αυτό. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τελευταίας συζήτηση που είχαμε στην Ολομέλεια για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Και μας είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί πλέον σκόπιμη την ενεργοποίηση του μηχανισμού κράτους δικαίου. Πώς έχει λοιπόν η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών της σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την πληρέστατη παρουσίασή σας των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα όσον αφορά το έκρης, είπατε ότι θα επιταχυνθεί η προσπάθεια για τη νέα μορφή του έκρης. Ποιο χρονοδιάγραμμα έχετε. Δεύτερη ερώτηση. Για τους ασφαλείς λιμένες. Ποιο είναι το δυσχερέστερο σημείο για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τον ασφαλή λιμένα με τη ΣΥΠΑ Και κάτι σχετικό. Το δεύτερο ενδεχόμενο για να αποφυφθεί η εμπλοκή πριν το τέλος του Ιανουαρίου. Διότι η ομάδα του Άθρου 29 είπε ότι έχουμε χρόνο μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις και για τη ροή των πληροφοριών. τίτη ερώτηση Ο Τίμωθη Κύρκοπ έκανε μια, πρόταση για την εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου, για το GDPR. Πρέπει να ξεκινήσει το έργο όσον αφορά την εφαρμογή, διότι η ποιότητα του GDPR εξαρτάται από την καλή εφαρμογή για τον κανονισμό ή την προστασία των δεδομένων. Είναι κάτι που είναι σημαντικό και για τα κράτη-μέλη. Εξετάζει την κατάσταση στην Πολωνία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς ξεκίνησαν να εμφανίζονται κάποια νέα φαινόμενα που παραβιάζουν τους κανόνες της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου και σταδιακά θα είναι σημαντικό να το θέσουμε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους συναδέλφους μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπόνη. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θα ρωτούσα για τον ασφαλή λιμένα. Πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Σίπελ και ο κύριος Μπόνι, να πω κι εγώ κάτι, μια ερώτηση. Αναφέρατε, αναφερθήκατε στις συναντήσεις που είχατε στη ΣΥΠΑ. Όταν προέκυψαν τα θέματα της τρομοκρατίας και είπατε ότι αυτά που συνέβησαν ε, δυσκόλεψαν τις συζητήσεις. Πολλοί συνάδελφοι στην Επιτροπή ασχολούνται με τον ασφαλή λιμένα και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Κάποια εικόνα μπορείτε να μας δώσετε. Πότε μπορούν να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ. Έγινε κάποια διακοπή. Πότε θα υποβληθεί η νέα πρόταση. Ξέρουμε ότι είναι περιπλοκότατο ζήτημα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα όμως. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και άλλος συνάδελφος. Η Σοράγια θέλει να πάρει το λόγο. Η Σοράγια Πόστ. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, Κυρία Γιώροβα, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Έχω τρεις ερωτήσεις να θέσω. Πρώτη ερώτηση που αφορά αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αναφερθήκατε στην προστασία της σεξουαλικής ταυτότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Δεύτερη ερώτηση. τα συναισθήματα κατά των τζιγκάνων, η, κατάσταση, η ατμόσφαιρα κατά των τζιγκάνων θα φροντίσει για την προστασία των Ρωμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ενταχθεί σε μια στρατηγική, εθνική, η καταπολέμηση αυτών των ανητικών συναισθημάτων. Τρίτον, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εντόπιση κάποιων εγκλημάτων που οφείλονται σε μυσαλλοδοξία. Ευχαριστώ, Σωράγια. Συναδελφοί, άλλο τίποτα. No. Um, but again, I think, and again. Και πάλι, κύριε Πίτροπε, σας είπα, είναι ένα συνήθιστο πρωινό σήμερα. Είχαμε μεγάλη ψηφοφορία και κάποια προβλήματα οργανωτικά και την Πέμπτη κάποιοι συνάδελφοι αποχωρούν νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη. Και ζητώ συγγνώμη και από τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Τουλάχιστον οι παρόντες είχαν περισσότερο χρόνο να επεκταθούν σε ερωτήσεις, που είναι μια μικρή πολυτέλεια που συνήθως δεν έχουμε. Και εσείς επίσης. Δεν θα σας πιέσω για αλλαγή. Βέρα, παρακαλώ με την ησυχία σας. Να απαντήσετε χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάτι να πεις για να μιλάς. Να πείτε ό,τι θέλετε, να σας πιέσω εγώ δεν θέλω. Και όποτε έρχεστε, ε, ο χρόνος είναι πάντα πάρα πολύ πιεσμένος. Και πάρα πολλές ερωτήσεις και πρέπει να τρέχετε για απαντάτε. Σήμερα είναι κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, αν έχουμε πολύ χρόνο, που όντως είναι τέλεια θα μπορούσαμε να έχουμε και ερωταπαντήσεις. Διάλογος δεν είπαμε ότι είναι. Και ε, συμπληρωματικές, αν έχετε παρακαλώ μην διστάσετε. Ναι. Μπορεί να με, και να με επικρίνετε από τις απαντήσεις που θα δώσω και να γεννηθούν και άλλες ερωτήσεις. Θέλω να απαντήσω πρώτα σε αυτό που είπε ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Uh, ότι έρχομαι και συζητώ μαζί σας. Είναι ε, καθήκον μου, μόνο. Εγώ λογοδοτώ στο Κοινοβούλιο και έχω τέσσερις επιτροπές στις οποίες λογοδοτώ αλλά η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, Πολιτικών Ελευθεριών ασχολείται με θέματα πάρα πολύ δύσκολα και ε, πάρα πολύ απαιτητικέ προκλήσεις. Ε, σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι καιροί. Είναι πάρα πολύ χαλεπή. Είναι πολλές οι κρίσεις εκτός της Ένωσης που δεν έχουμε εμείς πλήρη εξουσία για να τις λύσουμε, ούτε αρμοδιότητα. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε ευφυείς πολιτικές συνόρων, να ελαχιστοποιήσουμε τις ανητικές συνέπειες στην Ευρώπη, αλλά έχουν και πολλά προβλήματα στο εσωτερικό μας. Και αυτά θα πρέπει εδώ να συζητούμε. Και ένα από τα βασικότερα ερωτήματα είναι η σύγκρουση βασικών αρχών. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην ασφάλεια. Αυτό είναι στον πυρήνα του ασφαλούς λιμένα και όλων των άλλων συζητήσεων για την προστασία των δεδομένων και για άλλες πολιτικές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ερώτημα αυτό και κέριο. Πώς θα σταματήσουμε την αυξανόμενη μη σαλλοδοξία στην κοινωνία μας. Γιατί ζούμε ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα. Φεύγουν οι Εβραίοι από την Ευρώπη διότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στην Ήπειρό μας. Είδα και τα στοιχεία. Πόσοι έχουν εγκαταλείψει τη Γαλλία. βλέπουμε ένα τραγικό, ένα τρομακτικό φαινόμενο ε, λόγων μίσους σε όλη ε, την ε, κυβερνόσφαιρα. Το ίντερνετ εντάξει είναι τέλειο, φανταστικό και βοηθάει τον κόσμο, αλλά ο κυβερνοχώρος τώρα χρησιμοποιείται για τέτοιες κατακρίσεις και για τέτοιους ε, τρομακτικούς ιδεχθείς σκοπούς εγκλήματα μίσους, βία, λόγους, κηρύγματα μίσους. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ε, στεναροί και να τραβήξουμε μια γραμμή διαχωριστική ξεκάθαρη. Άλλο πράγμα είναι η ελευθερία της έκφρασης που θα πρέπει να είναι όσο γίνεται ευρύτερη, αλλά υπάρχει και ανάγκη δράσης δεν μπορεί να υποδαβλίζεις το μίσος και να καλείς εγκλήματα μίσους και ε, τα λοιπά. Αυτά θα πρέπει να σβήνονται, να διαγράφονται, να κατεβαίνουν από το διαδίκτυο. Όλοι προβληματιζόμαστε μέσα μας, αλλά... Κοιτάξτε, ας πούμε, το δικαίωμα στην ασφάλεια και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αν το συζητήσουμε δύο-τρεις, ο καθένας θα έχει ε, εσωτερικά άλλη αίσθηση και σε λίγο μπορεί και να τσακωθούμε. Δηλαδή φανταστείτε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για αυτό το θέμα που είναι τόσο προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες κόκκινες γραμμές να τραβήξουμε. Πολύ ε, άχαρο και δύσκολο αυτό το έργο, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τα χτυπήματα. Φανταστείτε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε και, επιπλέον και με τους Αμερικανούς, όχι μόνο μεταξύ μας, που έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι εστί ασφάλεια και τι ιδιωτική ζωή τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το πώς βλέπουν τα πράγματα. Αυτό τα λέω σε σχέση με το Safe Harbor, τον ασφαλή λιμένα. Ναι, κύριε Λόπε Αγγιλά, χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον σα, γιατί πραγματικά έχω ανάγκη να ακούω τι απόψει σα, εσά που ασχολείστε με όλα αυτά τα δύσκολα θέματα και εστιάζετε σε αυτά. Γιατί πρέπει να παίρνουμε δύσκολε αποφάσει, αλλά όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να είναι συλλογική αυτή η προσπάθεια. για να παίρνουμε κάθε φορά τη σωστή απόφαση. Σε αυτούς τους καιρούς που είναι πολύ απαιτητικοί επαναλαμβάνω και ξέρουμε ότι δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Μια και έξω πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις από την αρχή. Αυτούς τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Συγγνώμη που μακρύγορο Έφεγα όλο μου το χρόνο που είχα το απόθεμα. Να απαντήσω τώρα σε ερώτησή σας. Σε ερωτή σας. Έχετε, έχετε χρόνο. Λοιπόν, έπρεπε να ξεκινήσω από αυτή την εισαγωγική παρατήρηση για να σας πω πόσο σημαντικός είναι για μένα αυτός ο διάλογος. Με ευχαριστήσατε που ήρθα. Εγώ σας ευχαριστώ που έχω αυτή την ευκαιρία και οι ε, συνεργάτες μου, το επιτελείο μου που εργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα. Η κυρία Σίπελ ρώτησε κάτι για τη Eurojust. Μάλιστα είναι έργο αυτό και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δικό μου να είμαι σε μόνιμη επαφή με τον πρόεδρο της Eurojust και να κοιτούμε ε, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα και να αξιοποιούμε στο επακρό αυτό τον οργανισμό. Διεθνή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, και με τις τρίτες χώρες, τα Δυτικά Βαλκάνια, χώρες Μέσα Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, αλλά και με την Τουρκία, που θα πρέπει να συμμετέχει είναι κρίσιμο. Οι γειτονικέ μας χώρες, οι όμορες, θα πρέπει να καταπολεμούν το οργανωμένο έγκλημα με τρόπο αποτελεσματικό. Γιατί αν δεν πετυχαίνουν εκείνες, αυτό ε, επηρεάζει και τη δική μας ασφάλεια. Βεβαίω να ενισχυθεί η Eurojust, υπάρχουν ήδη κάποιες βελτιώσεις που παρατηρούνται και αύξηση του προϋπολογισμού αλλά και των ανθρωπίνων πόρων τους προβλέπεται για το 2016 και θα πρέπει να συνεχιστεί. Για το, γραφείο του Ευρωπαίου Σαγγελέα έκαναν ερωτήσεις και η κυρία Σίπελ αλλά και ο κύριος Κέρκοπ. Θα απαντήσω από κοινού λοιπόν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το εξή. Οι προεδρίες διαδέχονται μία την άλλη και ε, οι εξελίξεις αλλά δεν αλλάζουν οι αρμοδιότητες. Τελικά θα πρέπει να έχουμε ένα θεσμό ισχυρό. Δεν μπορεί να είναι αδύναμος, ε, ανίσχυρος και δεπανηρός. Τι να τον κάνουμε ε, τέτοιο γραφείο εισαγγελέα. Και το επαναλαμβάνω κάθε φορά στο Συμβούλιο, γιατί αυτή η αποδυνάμωση ε, των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων το ροκάνισμα αυτό, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο κόβω με μικρές τροπολογίες, ε, τελικά θα είναι τελείως αποστεωμένο αυτό το γραφείο και δεν θα έχει κανένα νόημα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν να δημιουργηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή εισαγγελία. Θέλουν να διατηρηθεί και ένας εθνικός σύνδεσμος. Αυτό το ζητούσε παγίως η κυρία Μακοβέη. το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα πρέπει να είναι ισχυρό, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Δεν χρειάζεται να είναι καμία τεράστια μηχανή, κανένας μηχανισμός που να μπαίνει ε, στη, σε ποινικέ διώξεις και να κρατάει τους υπόπτους 10 χρόνια γιατί με την πρόφαση ότι πρέπει να μεταφράζονται οι δικογραφίες ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία που να είναι συνεκτική, συνεπής και να είναι μια ομπρέλα των εθνικών ποινικών διαδικασιών ε, και διώξεων. Διότι πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο ε, χωρίς να θίγουμε ε, το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών και το δίκαιο ποινική δικονομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, γιατί τα συστήματα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν ανακριτές, ας πούμε. Υπάρχουν συστήματα που δεν έχουν ανακριτές. Έχουν άλλες δομές, ειδικέ και ειδικά μέτρα για τη δίωξη και τη διεξαγωγή της έρευνας και της ανάκρισης, δικονομικά δικαιώματα κτλ. Αλλά Υπάρχει μια ειδικότητα που είναι οι συναλλαγές. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουμε στην Ευρώπη. Υπάρχει μια μέθοδος για κάποια παραπτώματα ή πλημελήματα ε, που μπορεί κάποιος να πληρώσει και να σταματήσει η δίωξη. Και ο, ο καθηγητής ποινικού δικαίου αυτό το ονόμαζε ιδιωτικοποίηση της ποινική δικαιοσύνης σε κάποια ε, κράτη-μέλη υπάρχει δυνατότητα να εξαγοράσεις ε, ένα ποινικά κολάσιμο δίκημα πριν ε, διωχθείς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πως δυσκολίες να συγκρίνουμε τα συστήματα. Είναι πολύ διαφορετική η διαδικασία από χώρα σε χώρα. θα συμφωνήσουμε. Εκκρεμεί το άρθρο 216 γιατί στη Σλοβενία και την Πορτογαλία υπάρχουν ε, συνταγματικής φύσης προβλήματα. Διότι οι ανακριτές είναι ανεξάρτητοι, δεν μπορούν να δέχονται εντολές από κανέναν, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα δίνει εντολές στους ε, ανακριτές και στις διοκτικές αρχές των κρατών μελών. Άρα βλέπετε ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση, μπορεί να είναι λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε το συνολικό μοντέλο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και να είναι μια δομή αρκετά ισχυρή και με αρμοδιότητες. Ε, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών τα ακούσαμε, χορτάσαμε Ακούσαμε κάποιους υπουργούς που θέλανε να αποδυναμώσουν και να αφαιρέσουν αρμοδιότητες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Πάντως, στο Συμβούλιο εξακολουθώ να βλέπω ισχυρή υποστήριξη για τη δημιουργία ενός τέτοιου φορέα, του χρόνου συγκεκριμένα. να υπάρχει ένα γραφείο Ευρωπαίου Εισαγγελέα ισχυρό και να καταπολεμά τα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχομαι εδώ σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για το ΦΠΑ. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία ε, κατά της απάτης και οι απάτες στο ΦΠΑ θα πρέπει να καλύπτονται φυσικά ε, και, από και να διερευνώνται και να διώκονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είμαι 100% περισμένη. Μας βοήθησε και μια σχετική υπόθεση. Τώρα το Συμβούλιο τι λέει. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί και πάλι έχουμε να κάνουμε τις αρμοδιότητες των Υπουργών. Γιατί ξέρετε ότι αυτό το συζητούμε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη. Αλλά έρχονται και μα λένε οι Υπουργοί Δικαιοσύνη ότι αυτό είναι θέμα των Υπουργών Οικονομικών. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα. Ορισμένοι λέγουν ότι δεν μπορούν να τσακωθούν και με τον Υπουργό Οικονομικών του. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Προσπαθούμε να πείσουμε τους Υπουργούς Δικαιοσύνης να συμπεριληφθεί το ΦΠΑ η τελευταία συζήτηση ήταν πάρα πολύ σύντομη την Πέμπτη ή την Παρασκευή, πότε ήταν το Συμβούλιο, την περασμένη εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει. Το θίξαμε κάπως, έτσι, γενικά κάναμε μια σύνοψη στο που βρισκόμαστε και συμφωνήσαμε να φέρουμε τα στοιχεία με οριακές τιμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ε, ποια ε, ε, αδικήματα θα ε, διερευνά. Θα δούμε τις ποινικέ στατιστικές, γιατί τι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που έχουμε. Αν βάλουμε το όριο στις 100.000 ευρώ για σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα στο ΦΠΑ, θα κατακλειστεί η εισαγγελία από υποθέσεις. Θα πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη ε, για τις ποινικέ διώξεις για το ΦΠΑ και πόσο θα επιβαρύνει αυτό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να δούμε τις τάξεις μεγέθους δηλαδή. Εγώ ποια τακτική έχω. Καταρχάς να δούμε τα διασυνοριακά αυτά, τη σοβαρή εγκληματικότητα, την οργανωμένη στο ΦΠΑ και στην ε, καταπάτηση, μάλλον δίωξη της απάτης. Οι Ολλανδοί είπαν ότι θα το κοιτάξουν, βέβαια είναι δύσκολη η κατάσταση. Στο Συμβούλιο είπαμε, αλλά έχω συμφανίσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνη της ε, Ολλανδίας ότι την επόμενη φορά θα έρθουμε με στοιχεία για να μπορέσουμε να μπούμε σε πιο ρεαλιστικές ε, συζητήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και το ΦΠΑ. Έρχομαι τώρα στο Safe Harbor. Ακούσαμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Σίπελ. Ρωτήσατε για τη συνεργασία σε θέματα ποινική δικαιοσύνη. Ε, μεγάλο ζήτημα αυτό για το επόμενο έτος. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί πιο πολύ ψηφιακή ε, ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να είναι πιο γρήγορη η ανταλλαγή αυτή μεταξύ των σχετικών αρχών στα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιούμε τώρα ε, αμοιβαία νομική, νομική αρρωγή. Είναι ε, δύσκολο, βαρύ εργαλείο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη τεχνολογία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι στην επικοινωνία μα μεταξύ κρατών μελών. Και αυτό ήταν και το θέμα που διαπραγματεύτηκα και με τη Λορταλίν τη ΕΠΑ το ίδιο συζητήσαμε, ότι χρειάζεται να είναι πιο γοργή η ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ποινική δικαιοσύνη και γενικότερα σε θέματα δικαιοσύνη. Για τον ασφαλή λιμένα, το safe harbor, το θέμα του πώς θα ελεγχθούν ε, οι όροι αν πληρούνται το χρονικό πλαίσιο το οποίο ανέφερε και ο Κλοντ Μωράης. Είναι δύσκολη η υπόθεση αυτή. Και ομολογώ ότι σε θέματα προστασίας δεδομένων, όπως είπα και ευθύς εξ αρχής, καλούμαστε να κρίνουμε μεταξύ δύο αρχών, να βρούμε την ισορροπία μεταξύ προστασίας δεδομένων και ασφάλειας. Για τον ασφαλή λιμένα προτιστήθεται και μία τρίτη διάσταση, οικονομική πτυχή, και άρα σχηματίζεται ένα τρίγωνο. Νομίζω η κυρία Κορατσαμπίλτ έθεσε το θέμα των επιχειρήσεων και της νομικής αβεβαιότητας μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολη αυτή η άσκηση. Από τις συνομιλίες μου στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να πω ότι επέστρεψα με ένα αίσθημα επιτυχίας, ότι υπάρχει η ίδια αίσθηση κατεπήγοντος, ότι θα πρέπει πραγματικά να αντιδράσουμε γρήγορα. Ήμουνα επίση εντελώ ξεκάθαρη, όπου κι αν ε, συνομίλησα, ότι εάν πρόκειται να υπάρξει ένα καινούριο safe harbor, θα είναι μονομερή απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα το προτείνω αυτό στο σώμα των επιτρόπων, χωρί να είμαι βέβαιη ότι θα μπορώ να εφαρμόσω το σύστημα που ονομάζω Trust and Check. Εμπιστοσύνη και έλεγχος, κοιτώντας την ε, νομική αρχή και τις, ε, τα διατάγματα, τα προεδρικά στην Αμερική κτλ. Αν προσπαθήσει κανείς να αξιολογήσει κατά πόσον αυτή η ένωμη τάξη παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας όπως απαιτεί το δικαστήριο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ας περιμένουμε να αλλάξει η αμερικανική νομοθεσία προκειμένου να υπάρχει 100% βεβαιότητα για το τι μπορεί να κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος, τέτοια επιλογή. Εργαζόμαστε βάσει ενός συστήματος εμπιστοσύνης και ελέγχου. Πρέπει να υπάρχει και μια κάποια εμπιστοσύνη προς την Αμερικανική κυβέρνηση. Και για να σας δώσω κάποιο πιο συγκεκριμένα παραδείγματα διαπραγματευόμαστε με την, το Υπουργείο Εμπορίου και την ε, Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου στην Αμερική και με την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. Και θέσαμε τέσσερα σημεία και πριν μεταβούμε στην Ουάσιγκτον και ήθελα να το γνωρίζουν αυτό οι ομόλογοι μας στην Ουάσιγκτον, να ξέρουν ποιες είναι οι απαιτήσει μα, οι αξιώσει μα. Άρα είχα ανακοινώσει ότι θα διαπραγματευόμασταν τέσσερα σημεία. Καταρχά, τη μορφή τη δέσμευση τη επιστολή από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, ένα μνημόνιο κατανόησης ενδεχομένως. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε περαιτέρω. Στη συνέχεια, ζήτησα από τους αρμόδιους σε θέματα εθνικής ασφάλειας να μας δώσουν πιο ακριβείς ορισμούς για τις περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που, υπό τις οποίες ε, οι εθνικές αρχές, οι αμερικανικές αρχές ε, μυστικές υπηρεσίες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τις εταιρείες στα πλαίσια του Safe Harbor και η περιγραφή που μας έδωσαν δεν μας επαρκεί. Ήμουν σαφής για αυτό ότι θα πρέπει να ορίσουμε με πιο δεσμευτικό τρόπο αρχές και όρους όπως ε, η εθνική ασφάλεια. Τι είναι η εθνική ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Και αυτό θα μας, εδώ θα μας απαντήσουν οι Αμερικανοί ομολογοί μας αύριο. Έχουμε τεχνικές συζητήσεις αύριο. Και βάσει λοιπόν των συγκεκριμένων ορισμών σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις και τους συγκεκριμένους όρους, θα πρέπει να βρούμε και αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου. Γι' αυτό μίλησα για trust and check, εμπιστοσύνη αλλά και έλεγχος. Και θα συνεχίσουμε διαρκώς να ελέγχουμε. Υπό τη μορφή εκθέσεων από πλευράς ε, των Αμερικανικών αρχών για τον αριθμό των ετοιμάτων θα υπάρξει επανέλεγχος και επιβεβαίωση από πλευρά των επιχειρήσεων. Αυτό φυσικά δεν επαρκεί από μόνο του. Και ήθελα με κάποιο τρόπο να έχω πρόσβαση σε πιο εμπιστευτικές πληροφορίες. Αλλά αυτό φαίνεται να είναι αδύνατον. Τουλάχιστον όμως με τις εκθέσεις αυτές θα έχουμε κάποιες πληροφορίες για την τάση και θα ελέγξουμε και από πλευρά των επιχειρήσεων τι γίνεται ω μια βασική πηγή πληροφοριών. Αυτό που δήλωσα όμω επίσης προς τους Αμερικανούς ομολόγους είναι ότι θα ελέγχουμε και θα παρακολουθούμε και τη συνολική κατάσταση στην, στην Αμερική. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εταιρείε Safe Harbor, θα εξετάζουμε και τα μέσα ενημέρωση, θα μα πληροφορεί και η κοινωνία των πολιτών. Θα λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία των ε, whistleblowers. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και θα είμαστε σε διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης της κατάστασης. Αυτό ενδεχομένω να θεωρείται ότι είναι μια δύναμη πηγή πληροφοριών, αλλά συνδυάζει πολλές διαφορετικές οδούς και αυτό θα σχηματίσει μια συνολική εικόνα και την ε, ρήτρα αναστολής Αν ε, λοιπόν ε, λάβουμε επαρκείς ενδείξεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή θα ανασταλούν οι συμφωνίες αυτές. Αυτό για την πτυχή της παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο μηχανισμός αυτός με τις Αμερικανικές Αρχές για να εφαρμοστούν και όλα αυτά στην έκθεση. Το τέταρτο σημείο είναι και το πιο δύσκολο. Το πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης θα έχει στη διάθεσή του ενισχυμένα ένομα μέσα, σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει την ιδιωτική του σφαίρα, τα δικαιώματά του και τονίζω το ότι μιλάμε για ενισχυμένα νομικά μέσα, γιατί τα απλά νομικά μέσα δεν αρκούν. Θα πρέπει να είναι επαρκή τα ένεμα αυτά μέσα για να προστατεύσουν τον πολίτη. Αυτό λοιπόν το θέμα εξετάζουμε τώρα γιατί περιλαμβάνει τις ε, Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου από πλευρά της Αμερικής. Αυτό λοιπόν είναι το πιο δύσκολο ζήτημα γιατί πρέπει να εξεταστούν και θέματα δικαιοδοσίας. Ε, οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν, εξουσία, δεν έχουν δικαιοδοσία για τις ε, επιχειρήσεις που εισήγαγαν τα στοιχεία αυτά στις ΕΠΑ. Και λυπάμαι αν επισέρχομαι σε υπερβολικό βαθμό λεπτομέρειας, αλλά νομίζω ότι πολλοί από εσάς ε, γνωρίζετε το θέμα αυτό σε μεγάλο βάθος και ενδεχομένως να χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες. Το θέμα αυτό λοιπόν της εφαρμογής είναι το σημείο εισόδου για τα υπόλοιπα τρία. Γι' αυτό ξεχνά, ξεκινάμε λοιπόν από την κατάρτιση και την κατάστρωση του σημείου αυτού και το θέμα των ε, ένωμων μέσων. Χρονικός ορίζοντας τώρα. Διαρκώς ε, είμαστε σε διαρκή Αμα δουλεύουμε ακούραστα για το θέμα αυτό. Δεν θα πω και νυχθημερών, θα κάνουμε και Χριστούγεννα, αλλά το έχω ξεκαθαρίσει αυτό και στους συναδέλφους μου, ότι θέλω να δω τα κείμενα, τα κείμενα μπροστά μου, τα κείμενα με τις δεσμεύσει από πλευράς των Αμερικανών, τις αποφάσεις και όλα αυτά τα κείμενα για το μοντέλο εφαρμογής. Μέχρι το τέλη του Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει κατά πόσον το Safe Harbor θα ξαναλειτουργήσει ή όχι. Το καινούριο Safe Harbor και θα πρέπει να το βρούμε και ένα καινούριο όνομα, να το ξαναβαφτίσουμε. Και πάλι λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι είναι δικαίωμά μας να πάρουμε τις ε, απαραίτητες αποφάσεις. Δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει οδηγία που προβλέπει τη μεταφορά σε τρίτες χώρες. Και παρέχει κάποια σχετικά εργαλεία. Αυτά είναι τα εργαλεία με τα οποία τα οποία παρήχαμε στις εταιρείε με την ανακοίνωσή μου στις 6 Νοεμβρίου. Δεν είναι λοιπόν έκτακτα αυτά τα εργαλεία, αυτά τα μέσα, είναι τα τακτικά, προβλεπόμενα εργαλεία μέσα για τις μεταφορές προς τις χώρες. Τα επιπλέον εργαλεία επίσης, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την αυστηρή εποπτεία των ε, αρμόδιων για την προστασία των δεδομένων αν δεν υπάρχει επαρκή προστασία. Επαρκής προστασία. Όπως ε, μετά την απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει ότι συμβαίνει στην Αμερική. Αν δούμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η μεταφορά τέτοιων δεδομένων και πόσο η οικονομία και οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων, αυτό μας εξωθεί στην κατάρτιση ενός ειδικού ενός καθεστώτος ε, που θα επιτρέπει τη μεταβίβαση αυτή δεδομένων με τη σωστή προστασία από Αμερικανική πλευρά. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αν δεν υπάρχει η κατάλληλη προστασία από την αμερικανική πλευρά. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιο χρόνο ακόμα, αλλά και ο χρονικός ορίζοντας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι κατάλληλη προθεσμία ο Ιανουάριος. Είναι άλλωστε και η καταληκτική ημερομηνία που έχουν θέσει και οι υπόπτες ε, προσωπικών δεδομένων που έχουν ε, πει ότι από την ημερομηνία αυτή και μετά θα εφαρμόσουν τα εργαλεία της οδηγίας. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ολοκληρώσουμε το καινούργιο αυτό πλαίσιο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Και πιστέψτε με, έχω δαπανίσει μεγάλο κομμάτι του πολιτικού μου κεφαλαίου προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαι και παλιωμοδίτησα, ξέρετε, είναι σχεδόν θέμα τιμής αυτό πλέον για μένα. Αλλά εκ παραλλήλου αποτελεί και ένα θέμα τεράστια σημασία για τι επιχειρήσει και το οποίο προωθούμε από πλευρά ε, Ευρώπη και Αμερική νύχθη ημερών. Λοιπόν, θα ήθελα να δω Μήπως υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Σωράγια, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Γρήγορα, γρήγορα, σε παρακαλώ. Α, είχε... Α ήθελες να... ήθελατε να πείτε κι άλλα. Δε. Λοιπόν, ήθελα... The, yeah. the safe harbour because there were many, uh, many, many questions. Just, just, just because one colleague you wanted to ask a question as that. Λοιπόν, Ήθελα απλώς να ακούσω κάποιον που μη τυχόν είχε μείνει απ' έξω. Αν μπορούμε να ακούσουμε την ερώτηση της Οράγιας πρώτα και μετά συνεχίζετε. Λοιπόν, ήθελα μία από τις ερωτήσεις που είχα θέσει πριν να θέσω ξανά. Η απόφαση πλαίσιο για τα, τα, τα εγκλήματα μυσαλλοδοξίας. Τι γίνεται εκεί. Υπάρχει απόφαση πλαίσιο για τα εγκλήματα μυσαλλοδοξίας Μήπως πρέπει να διευρυνθεί για να καλυφθούν και άλλες πτυχές. Είπατε ότι δεν είναι δυνατόν σαν απάντηση μπορείτε να μας πείτε όμως ποια είναι η κατάσταση που βρισκόμαστε. Θα μπορούσαμε να έχουμε λεπτομερέστερη απάντηση όσον αφορά τη θέση σας επ' αυτού. Διότι είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αφορά μια κατηγορία τόμων που εκτίθενται σε αυτού του είδους τα εγκλήματα. Είναι συμπληρωματική ερώτηση αυτές που είχα θέσει πριν. Η Επίτροπος νομίζω ότι θα ήθελα να το θίξει. Τζούντι, θες να ρωτήσει κάτι. Όχι. Νόμιζα ότι τελείωσε. Θα περιμένω μέχρι να τελειώσει. Γιατί είναι ένα ερώτημα που αφορά τους Λουάδ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που διακόψα σε λάθος σημείο, κύριε Επίτροπε. Άλλος της αγορεύειν βούλετε; Επίτροπε. Συνεχίστε. Συγγνώμη που μακρηγορώ. Μακρηγόρησα για τον ασφαλή λιμένα, αλλά βλέπετε ότι είμαι kind of a to... Ε, λοιπόν, είναι θεραπεία. Με πλημμυρίζει. Στα αγγλικά δεν το λέμε αυτό. Αυτό που είπατε, full of it, σημαίνει κάτι άλλο. Είμαι πολύ ενθουσιώδης, θα πρέπει να πείτε. Μην λέτε full of it. Σημαίνει, λέει ο Πρόεδρος, κάτι αρκετά διαφορετικό. Έχουμε αρκετό χρόνο, οπότε δεν έφαγα πρωινό και δεν είμαι γεμάτη από κάτι άλλο είσαστε πολλά πράγματα, αλλά όχι full of it, λέει χαριτολογώντα ο πρόεδρο. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στα σοβαρά θέματα. Έχουμε νομοθέτημα το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσει το θέμα της ασφαλείας Έχουμε πρώτα απ' όλα την απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πρέπει να το εξετάσω αυτό, διότι καλύπτει κάθε είδους ε, ομιλίες μίσους, μυσαλλοδοξίας που μπορεί να παροτρύνει σε εγκλήματα ε, και βία. Και τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν το μέτρο σωστά, να το εφαρμόσουν. Πρέπει να ελέγξω την κατάσταση για τους ΛΟΑΔ σίγουρα αντιτσιγανισμός, αντισημιτισμός, Ισλαμοφοβία, ε, όλα αυτά τα πράγματα καλύπτονται και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι έτοιμα να κινηθούν και αφορούν θέματα ποινική δικαιοσύνης. Υπάρχει κάτι, έπρεπε να έχει εφαρμοστεί τα 16 από τα 28 κράτη-μέλη, υπάρχουν και κάποιες αυτοεξαιρέσεις opt-out, στα 16 κράτη-μέλη βλέπουμε έλλειψη καλής εφαρμογής της αποφάσεως πλαίσιο. Οπότε είμαστε σε επαφές με κάθε χώρα ξεχωριστά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στα πλαίσια συνεργασία με τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, για να μειωθεί και αυτού του είδους η έκφραση, η μυσαλλοδοξία και στο διαδίκτυο. Και καλό τα κράτη-μέλη και τους υπουργού σε κάθε συμβούλιο και μάλιστα στα τρία τελευταία συμβούλια να το εξετάσουν το θέμα διεξοδικότερα και να εφαρμόσουν σωστά την απόφαση πλαίσιο. Δεύτερον, η οδηγία μετά που έχουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Δεν θέσατε ερώτηση πάνω σε αυτό έτσι, όχι. κατάλογος δράσεων για τους ΛΟΑΔ. Ποια είναι η κατάσταση παρούσα. Γίνονται συζητήσεις. Γιατί να μην έχουμε σχέδιο δράσεως, γιατί να μην έχουμε στρατηγική. Το απολαμβάνω και αυτό στα πλαίσια της πολιτικής για την ισότητα των φύλων και για τα θέματα των φύλων. Έχουμε στρατηγική δέσμευση που έχουμε αναλάβει και κάποιο μα κατακρίνει διότι δεν έχουμε διαμορφώσει στρατηγική. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση. Αυτή εδώ είναι η δέσμευση. Είμαι επίτροπος υπεύθυνη για τον τομέα. Αν δείτε αυτή την ε, ανακοίνωση του έγγραφου αναλαμβάνονται δεσμεύσεις και άλλων γενικών διευθύνσεων. Εδώ είναι ή κάπου αλλού το έχουμε αυτό. Α, υγεία. για την εμπλοκή της Γενικής Διευθύνσεως Υγείας, ΣΑΝΚΟ. Αναφέρεται ότι άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται από αυτού, άλλες γενικές διευθύνσεις έχουν πλήρη επίγνωση του μερτικού τους της προσπάθειας, διότι και άλλοι συνάδελφοι συντάσσουν και αυτοί αυτό το έγγραφο είναι ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταστεί σαφές ότι είναι σημαντική πολιτική για μας. Κυρίως υπό το φως των προσφάτων γεγονότων θα γνωρίζετε ότι ΕΠΣΚΟ στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης περασμένης εβδομάδος δεν κατορθώσαμε να εγκρίνουμε την καταχωρημένη ε, σχέση ε, και την περιουσία ε, που τα δικαιώματα σαν αυτή την περιουσία λόγω γάμου και όλα αυτά η Πολωνία δεν μπορούσε να δεχθεί το, το, την προσέγγιση, υπήρχαν συνταγματικά κολλήματα για τη χώρα αυτή, όλα τα άλλα κράτη-μέλη είπαν πολύ γρήγορα ότι θέλουμε ε, ενισχυμένη συνεργασία και θα είμαστε όλοι συμμετέχοντες διότι για θέματα οικογενειακού δικαίου χρειαζόμαστε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία μέσω της διευρυμένης συνεργασίας. Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο δράσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει στα πλαίσια σχεδιασμού εν διαχειρίσεως και διάθεση στην αγορά ούτε ΣΥΠΗΝ. Είναι συλλογική προσπάθεια, είναι καλό το νομικό καθεστώς. Εδώ αναφέρουμε σαφώς τι θα κάνουμε. Και θέλουμε να συντάσσουμε αιτήσιες εκθέσεις πρόοδου όσον αφορά τα ζητήματα των ΛΟΑΔ. Η οδηγία για την ίση αντιμετώπιση, ίση μεταχείριση είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Είμαι απογοητευμένη διότι στα συμβούλια που συμμετείχα όλοι αναφερόταν στην αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιας νομοθεσίας διότι καλύπτει το κενό όσον αφορά την νομοθεσία κατά των διακρίσεων όμως υπάρχει πολύ μικρή προθυμία εγκρίσους διότι η οδηγία έμεσα έχει δημοσιονομικές συνέπειες διότι χρειάζεται, χρειάζονται μέτρα και κατασκευές για ανθρώπους με αναπηρία που κινούνται με αναπηρικά καροτσάκια. Ενημέρωσα ε, τους ε, υπουργούς για την πράξη, για το νομοθέτημα περί προσβασιμότητας που ίσως να αποτελεί μια λύση αλλά ακόμα δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική βούληση για έγκριση. Βασίζομαι πολύ στην Ολλανδική Προεδρία για αυτό το θέμα, διότι οι Ολλανδοί είναι πολύ καλή όσον αφορά αυτές τις πολιτικές, έτσι δεν είναι. Όχι. Πάει η αισιοδοξία σας, λέει ο Πρόεδρος. Όσον αφορά τα παιδιά, βρίσκω ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στις ε, σχετικές πολιτικές και τα παιδιά. Σχεδιάζω να κάνω δύο πράγματα. Παρόμοια με τον κατάλογο δράσεων για τους ΛΟΑΔ, Στη γενική μου διεύθυνση προγραμματίζω να κάνουμε παρόμοια πράγματα για τα παιδιά. Άρα θα έχουμε πλήρη κατάλογο δράσεων που θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση για τα παιδιά στην Ευρώπη. Σχεδιάζω και επεξεργάζομαι τους συναδέλφους κάτι βραχυπρόθεσμο. Η κατάσταση για τα συνόδευτα παιδιά και τα παιδιά μετανάστες είναι φρικτή. Όταν δοκίμασα τις γρήγορες λύσεις, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, ανακάλυψα ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις. Και αποφάσισα παρόλα αυτά να υποβάλω έναν κατάλογο δράσεων που θα πρέπει να δρομολογηθούν γρήγορα. Θα το υποβάλω αυτό το κείμενο στο σώμα των επιτρόπων. Θα υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία πόσα παιδιά έχουμε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τι απειλέ αντιμετωπίζουν, ποιου κινδύνου και ποια είναι τα καθήκοντα των σχετικών φορέων. Θα υπάρχουν τρία κεφάλαια για τα καθήκοντα, ένα κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα για τα κράτη-μέλη και το τρίτο για τις διάφορες οργανώσεις. Θέλω να συναντηθώ με εκπροσώπους των μεγάλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, των μεγάλων οργανώσεων που θα πρέπει κανονικά να βοηθήσουν την εξέβρεση λύσης, γιατί η κατάσταση είναι φρικτή σε αρκετά κράτη-μέλη. Αυτό είναι, αυτή είναι η γρήγορη λύση που θέλω να προωθήσω. Ελπίζω να καταφέρω να επιστήσω την προσοχή όλων των σημαντικών φορέων, ούτω ώστε κάτι να γίνει τώρα, αύριο. Λοιπόν, μεταρρύθμιση στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Υπάρχει μεγάλη πολιτική βούληση, αυτό διαισθάνομαι, για να ολοκληρωθούν οι τριμερείς διάλογοι. Υπάρχουν αρκετά δύσκολα σημεία προς επίλυση. Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να διευθετηθούν. Ένα είναι η, η, ε, εμπεριστατωμένη σύμφωνη γνώμη, ε, ενήμερη σύμφωνη γνώμη του υποκειμένου που αφορούν τα στοιχεία. Το θέμα των στοιχείων, αυτός που των στοιχείων είναι πάρα πολύ σχετικό. Είμαστε περήφανοι που θα έχουμε ομοιόμορφους κανόνες γι' αυτό, που θα πρέπει να εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη με ομοιόμορφο τρόπο. Αυτό δεν αφορά μόνο τη συμφωνία επί της χρήσεως των κυρώσεων, αλλά και πολλά άλλα θέματα όπου οι κανόνες δίνουν στις αρχές για την προστασία των δεδομένων διακριτική ευχέρεια. Επεξεργαζόμαστε εφαρμοστικές πράξεις, κατευθυντήριες γραμμές και θα γίνουν εκστρατείες κυρίως το 2017 απευθυνόμενες προς τις επιχειρήσεις και προς το κοινό περί της μεταρρυθμίσεως και τι της αφορά. Εάν θα μπορούσατε να κλείσετε διότι τελειώνει και ο χρόνος. Έχετε κάποια ερώτηση, περιμένατε μέχρι το τέλος. Ναι. Λοιπόν, γρήγορα παρακαλώ. Πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Σόγκορ, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μια σύντομη ερώτηση. Σήμερα το πρωί Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το σύστημα παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ποιες είναι οι δυνατότητες για ένα πλαίσιο ελέγχου. Υπάρχει μια σύμβαση ε, και αυτό που λέγεται ένα δημοκρατικό σκόρμπορκο, επίνακας επιδόσεων, ή βαθμολόγιο. Πώς βλέπετε και τις προοπτικές, υπάρχει τέτοια δυνατότητα να δημιουργηθεί τέτοιο είδους σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου. Επανειλημμένα έχω ρωτήσει ε, προκατόχου σας για τις εθνικές ε, μειονότητες που δεν είναι ούτε τσιγκάνοι, ούτε Ρωμά, ούτε παιδιά, ούτε μουσουλμάνοι, ούτε ε, μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Αλλά είναι μειονότητα γιατί είναι σε μία χώρα και μιλούν άλλη γλώσσα ή έχουν άλλη θρησκεία τουρκική μειονότητα στην ναι. Ελλάδα και στη Βουλγαρία, ουγγρική μειονότητα ε, στην Ρουμανία και τη Σλοβακία κτλ. Θα μας φύγει η διερμηνία, λέει ο πρόεδρος στις 12.30. Αν θες να απαντηθεί η ερώτησή σου. Σωραία, τρίτη φορά θα πάρεις το λόγο. Πάρα πολύ γρήγορα, θα φύγουν οι διερμηνείς. Eh, eh, ναι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν απαντήσατε στην ερώτησή μου, Βέρα. Έκανα μια ερώτηση που είχε να κάνει με τον αντιτσιγκανισμό, τα εχθρικά προς τους Ρωμά αισθήματα. Ε, υπάρχει μια στρατηγική σε σχέση με τις εθνικές στρατηγικές. Θα μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε. Υπάρχουν ιδιαίτερα ιδεχθεί και αποτρόπα εγκλήματα. Okay, so if, if, και θα μπορούσε να διευρυνθεί αυτό και με τους ΛΟΑΔ. Μπορείτε να απαντήσετε κύριε Επίτροπε σύντομα στα δύο ερωτήματα για να κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα. Θα το τσεκάρω. Αυτό το τελευταίο θα το ελέγξω. Όπως και στη στρατηγική τους Ρωμά και τις εθνικές στρατηγικές. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή όμως να αντιδράσω. Δεν ήθελα να αποφύγω το θέμα της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για το κράτος δικαίου, αλλά και αυτή η τελευταία ερώτηση ήταν στενά συνδεδεμένη. Ξέρω ότι το συζητήσατε με τη Βιβή Μίχου σήμερα το πρωί. Ελπίζω Αλλά πώς να το μετρήσεις αυτό με ποσοτικό τρόπο ή με πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Το κράτος δικαίου. Δεν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, η οικονομική πειθαρχία. Πώς μετριέται αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήμουν υπέρ ενός τέτοιου μηχανισμού, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Κατά πόσο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα μαγικό ραβδί. Ε, πρόσφατα μετέβαινε και στην Ουγγαρία γιατί ήθελα να δω ειδείς όμαση και να νιώσω την ατμόσφαιρα στη χώρα. Και εγώ προέρχομαι από μια χώρα και που έχω ζήσει το ε, ολοκληρωτισμό και έχω ένα αίσθηκτο έτσι τα πιάνω αυτά τα φαινόμενα και τις τάσεις που έχουν να κάνουν ε, με ολοκληρωτισμό και δεν το ένιωσα αυτό στην Ουγγαρία. Ξέρω τι κάνουν με την ομοθεσία τους και με το, ε, τις μήκαιο της και τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, κάτι πάει στραβά στη χώρα, αλλά ε, δεν θα πρέπει ε, αυτόματα αυτό να πούμε ότι είναι ένας μηχανισμός για το κράτος δικαίου και να πούμε ότι α, έχουμε πρόβλημα ή έχουμε την υποψία ότι συστηματικά και ε, διαρκώς παραβιάζεται η συνθήκη. Είναι με ένα άλμα αυτό. Χρειάζεται ίση μεταχείριση για τα κρατη και αντικειμενική αξιολόγηση. Αν υπάρχει τέτοιο μηχανισμό γιατί όχι, αλλά δεν τηρώ επαναλαμβάνω ότι είσαι μου. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά ε, για μένα και σας ευχαριστώ και με πολύ ενθουσιασμό προσβλέπω στο μέλλον. Βεβαίως και με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τα είπατε Βιέρα. Ιδιαίτερα όσοι μπήκατε στον κόπο να μείνετε, πρέπει να ξαναπώ ότι ήταν πολύ περίεργο το πρωινό σήμερα. Πολύ... Έχουν τη δυναμική τους οι συνεδριάσεις. Ευχαριστούμε την Επίτροπο που απάντησε με την ησυχία της και σε βάθος και σε ουσία. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά θέματα ε, την εισαγγελία, το ΛΟΑΔ, ε, πάντα ε, πολύ σημαντικά θέματα έχετε και χειρίζετε και δεν έχουμε πάντα την ευκαιρία να τα συζητούμε σε τέτοιο βάθος. Θα ήθελα λοιπόν να πω για το Safe Harbor ένα τελευταίο. για το χρονοδιάγραμμα, καθώς θα το ε, μάθουμε να μας ξανάρθετε στην αρχή του 2016 με τα η συνεδρίασή μας ε, για να έχουμε μια καλύτερη ιδέα πού το πάμε. Γιατί είναι κάπως επίγον. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για τη συνεδρίαση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Πολύ ουσιαστική συνεδρίαση και για τον ενθουσιασμό σας. Ευχαριστώ πολύ.